Αγαπητοί συναδελφοί, καλησπέρα σας και στο συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Το τρένο μου είχε καθυστέρησει φτάνοντας στις Βρυξέλλες. Είχα πει στην κυρία Φόρτ το μεταξύ ότι θα ήταν καλό να έρθει να αναλάβει τα ενία μέχρι να φτάσω. Έχουμε αργήσει κάπως. Ας ξεκινήσουμε. Αλλά πριν να ξεκινήσουμε, έχουν και πάλι οι διερμηνείς ζητήσει μία δήλωση για τις κινητοποιήσεις τους. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας για να ακούσετε στη γλώσσα σας τη δήλωση. Βρισκόμαστε στην 21η ημέρα κινητοποιήσεων διαμαρτυρία και η διοίκηση παραμένει αμετακίνητη. Αντιθέτω, μετά από 8 μήνε διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Προσωπικού, ο Γενικό Γραμματέα κλείνει τη στάση του. Για τη σημερινή συνεδρίαση δεν ε, έχουμε επιταχθεί, αλλά δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου. Σα ευχαριστούμε για την προσοχή σα. Okay, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ακούσαμε το, το μήνυμα, δεν θα υπάρξει υπέρβαση ωραρίου και θα τηρήσουμε βεβαίως αυτή τη τακτική. Ερωτώ αν έχετε παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Δεν μου έχει ζητηθεί τίποτα. Μπορούμε να την εγκρίνουμε λοιπόν. Μία ανακοίνωση έχω. Ευχάριστη. Καλωσορίζουμε νέο συνάδελφο νέα συνάδελφο. Η κυρία Βάιρνεν, όπως ξέρετε, έχει πάει. Ο κύριος Βάιρνεν έφυγε, πήγε στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Δεν είχα ενημερωθεί βέβαια πριν φύγει για να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Αλλά έχουμε την αντικαταστάτρια, την κυρία Μίριαμ Βέικάπερα, της οποία η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίριαμ, θες να πεις δύο λόγια στην Επιτροπή μας, παρακαλώ. Και καλώς ήρθες. Στα αγγλικά. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με χαρά είμαι εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που περνώ εδώ. Ουσιαστικά ανταλλάξαμε τις θέσεις μας με τον κύριο Βάιρου. Αν ήρθε εκείνο στο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και εγώ εδώ. Επί 11 χρόνια ήμουνα μέχρι τώρα ε, βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Φιλανδίας, άρα έχω ε, συμμετάσχει στα ογίγναστα για αρκετό καιρό, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Well, you're, very welcome and of course... Καλώς ήρθατε θέρμα. Θερμό καλώς όσμα βεβαίως ότι είναι δύσκολο ένα μόλις χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές με το τέλος της θητείας. Αυτό μου συνέβη και εμένα, ξέρετε. Είναι δύσκολο να μπει κανεί στη δουλειά όταν οι άλλοι όλοι γνωρίζονται μεταξύ του, έχουν κάνει τη δουλειά για χρόνια, μέχρι να γνωρίσει κανεί το προσωπικό κτλ. Αλλά να ξέρετε ότι είναι στη διάθεσή σα όλοι οι συνάδελφοι και το προσωπικό για οποιαδήποτε απορία έχετε. Με χαρά λοιπόν σα καλωσορίζουμε και πάλι. Προχωρώ στο σημείο 3, πρακτικά τη συνεδρία τη 24 η Απριλίου, κοινή με την Επιτροπή των Γυναικών, Δικαιωμάτων των Γυναικών. Αν έχετε κάποια σχόλια παρακαλώ στην γραμματεία μέχρι το τέλος συνεδρίασης ιδάλλως εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 4. Συντονιστές. Πρακτικά της 16ης Μαΐου και 19ης Ιουνίου το ίδιο ισχύει ότι σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης προς τη γραμματεία. Σημείο 5. Ανακοίνωση από την Επιτροπή. Έχει η Επιτροπή κάτι να μας ε, ανακοινώσει είτε από την ΔΕΦΚΟ είτε από την Ενκό, Ο Κάστερ Σόρενσεν πρώτος, από την ΔΕΦΚΟ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα για την ε, φάση μετά το κοτονού. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι στις 22 Ιουνίου, την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, έλαβε την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Συμβούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, με τις χώρες της Αφρικής Καραϊβικής και Ειρηνικού. Το περιμέναμε, έγινε και αυτή η ανάθεση εντολή και ξεκινούν οι συνομιλίες. μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, επομένως έχετε και την εντολή σας. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίω τι εξελίξει και το πώ θα αντικατοπτριστεί σε αυτές τι συνομιλίε το δικό μα ψήφισμα. Θα το συζητήσουμε σε μια από τι προσεχείς μα συνεδρίε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ για την ανακοίνωση και τώρα ο κύριο Λεφανσου από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Ναι, Wolfgang Streiter από την ΕΚΟ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και την παρουσίαση. Ε, πρόεδρε, θέλω να ενημερώσω κατόπιν της υπόσχεσης που είχε δώσει ο Επίτροπος ε, κατά τη διάρκεια του διαρθρωμένου διαλόγου το Μάιο, ότι τώρα έχει ξεκινήσει η πρόταση για την ε, εκπαίδευση και ιδιαίτερα με έμφαση στις περιοχές ε, που βρίσκονται σε κρίση για την υποστήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευση με βάση και το θεματολόγιο του 2030 για την εκπαίδευση. Έχουμε στην Επιτροπή τον, ε, επιλέξει τη διασύνδεση της, της εκπαίδευσης σε κάθε άλλη δραστηριότητα και κυρίως στην ανάπτυξη με τέσσερα κυρία θέματα, θεματικές ενότητες ε, συνεργασία με τους εταίρους για μια ταχεία και καινοτόμο εκπαίδευση και προσαρμογή. Δεύτερον, ε, συμπερίληψη ένταξη. Τρίτον, ειρήνη, προστασία. Και τέταρτον, ποιοτική εκπαίδευση για καλύτερο αποτέλεσμα της μάθησης της μαθησιακής διαδικασίας. Και για να κλείσω θα ήθελα να πω ότι θα έχουμε και τη σχετική χρηματοδότηση, όπως σας είπε και ο Επίτροπος το Μάιο. Εξασφαλίστηκε ένα ποσοστό 8% από, συνολικό μας, από τη συνολική μας πρικοδότηση φέτος για τις ε, περιοχές κρίσεως και την εκπαίδευση αυτές, του χρόνου θα γίνει 10%. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Βλέπετε δηλαδή ότι κάποια πολιτική μπορεί να αλλάζει, απλώς εδραιώνεται η πολιτική που ήδη υπάρχει. Ίσως πρέπει να καλέσουμε τον Επίτροπο να έρθει να μας μιλήσει. Κοιτάξτε, για εδραίωση πρόκειται και πρόκειται για ένα πρώτο ουσιαστικά έγγραφο πολιτικής ε, γραμμή από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της εκπαίδευση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε έκθεση για την εκπαίδευση στην αναπτυξιακή πολιτική και άρα πρέπει να τηρηθεί ενημέρωση και ο Επίτροπος ο εισηγητής και είμαι σίγουρη ότι και ο Επίτροπο Τηλιανίδη θα μπορέσει να έρθει να μα μιλήσει για αυτέ τι πολιτικέ γραμμέ και τι επιλογέ που οπωσδήποτε η Επιτροπή μα έχει υποστηρίξει επανελειμμένως τα τελευταία χρόνια. Σα ευχαριστώ πολύ και προχωρώ στο σημείο 6 τη θάσευση της παγκοσμιοποίησης, εμπορικές πτυχές. Σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή ΙΝΤΑ το Μάιο στις 17 Μαΐου δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφο αναλογισμού με τίτλο «Τη μάθευση της παγκοσμιοποίησης» και το Σεπτέμβριο του 2017 ε, δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Ισορροπημένη και προοδευτική πολιτική εμπορίου για την μάθευση της παγκοσμιοποίησης». Έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, ο κύριος Κριστιαν Πρέντα είχε αναλάβει τη γνωμοδότηση. Ο κύριος ε, Μπόγκαρτ είναι εδώ τώρα για να τον εκπροσωπήσει. Θα μιλήσω εκ μέρου του κυρίου Νταμπρέδα, ο οποίο δεν μπόρεσε να βρίσκεται στη σημερινή συνάντηση. Ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπόρεσε να εργαστεί σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και να παρουσιάσει το αρχικό σχέδιο τη γνωμοδότηση ε, τη Επιτροπή μα ε, στου συναδέλφου. Είναι σημαντική η τυθάσευση τη παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη, αλλά και για του εταίρου μα στι αναπτυσσόμενε χώρε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τις θετικά, τα θετικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης, αλλά τα αρνητικά. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και έχοντας υπόψη και τις δεσμεύσεις μας με, για τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Η αξιοποίηση της παγκοσμιοποίησης ε, είναι αναγκαιότητα δεδομένου ότι δεν καλύπτονται ε, επαρκώς όλες οι αναπτυξιακές ανάγκες εκεί. Ο ιδιωτικό τομέα παίζει σημαντικό ρόλο στην ε, χωρί αποκλεισμού και βιώσιμη ανάπτυξη. Το σχέδιο γνωμοδότηση που παρουσιάζουμε εδώ παρουσιάζει τη σταθερή θέση τη Επιτροπή μα ότι στα θέματα ανάπτυξη ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να δρά με τι κοινέ αξίε και τι ίδιε αρχέ ε, για αποτελεσματική επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, η γνωμοδότηση ε, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να, υλοποιήσει, να ενισχύσει τις πολιτικές της ε, για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνάδει αυτό με την ιδέα της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου του 2017 με τίτλο μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική για τη διθάσευση της ε, παγκοσμιοποίησης, για την πρόθεση των οικομενικών αξιών που υποστηρίζει και η Επιτροπή. Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία να υπάρχουν ολοκληρωμένες διατάξεις για κοινωνικά, ε, εργατικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, όπως και για τη βιώσιμη ε, ανάπτυξη. Να υπάρχουν τα σχετικά κεφάλαια δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν που είναι παγκόσμιο επίπεδου και που εμφανίζονται καθημερινά, πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιτύχουμε ένα χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Ο κύριος Πρέντα θέλει να υπενθυμίσει ότι μερικέ φορές έχουμε την τάση να βλέπουμε το εμπόριο και την ανάπτυξη ως αντικρώμενες δυνάμεις. Αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Το εμπόριο φυσικά δεν πρέπει να το βλέπουμε ως αυτό σκοπό αλλά κατά την άψη του εισηγητή ε, μια εμπορική πολιτική ελεύθερη χωρίς ε, αποκλεισμούς μπορεί να βοηθήσει την εκρίζωση της στόχιας. Επειδή είναι εισηγητή ε, τη Συνοχή Πολιτική για την Ανάπτυξη, ο κ. Πρέντα ήθελε να επιμείνει σε αυτή τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη του στόχου τη αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι αναπτυσσόμενες χώρε. Συνεπώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά να αξιολογεί την επίδραση των δικών τη εμπορικών πολιτικών στι τρίτε χώρε Δύο άλλα σημεία αναφέρονται στην γνωμοδότηση του κ. Πρέντα. Το πρώτο αναφέρεται στι οικονομικέ συμφωνίε εταιρική σχέση. Σημαντικό εργαλείο για την πρόθεση τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του εμπορίου εφόσον συνοδεύονται από τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα. Το δεύτερο σημείο, επίσης σημαντικό, ε, μια στροφή προς το μέλλον ε, με την ε, επέκταση, ε, με την διάδοση όλων των σχετικών τεχνολογιών και πολιτικών. Υπάρχει συμμετοχή του Επιτρόπου Γκαμπριέλ σε αναπτυξιακά αυτά θέματα και το υποστηρίζουμε αυτό μαζί και με τις περαιτέρω επενδύσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών παγκοσμίων. Ο κύριος Πρέντα προσβλέπει στη συνεργασία του με τους για βελτίωση του κειμένου και με πρόταση διαφορών τροπολογιών δεδομένου των περιορισμών χώρου ε, στην γνωμοδότηση κάποιε ιδέε χρειάστηκε να μένουν απ' έξω. Ο ίδιο έχει προτείνει κάποιε τροπολογίε για να εξεταστεί το ζήτημα τη φοροδιαφυγής στις εμπορικές εμπορικέ συμφωνίες. να υπάρχουν σχετικές διατάξεις, καθώς και τα προτιμησιακά σχέδια, καθώς και τα ε, επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Βρίσκονται εδώ κάποιοι σκιώδε εισηγητέ. Η Έλλης Λάιν πρώτη από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέντα. Ευχαριστούμε ε, κύριε Βέντα που μιλήσατε εκ μέρου ε, του κύριου Πρέντα για αυτή την πολύ σημαντική γνωμοδότηση η οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβει ισχυρή υποστήριξη. Η παγκοσμιοποίηση βοηθάει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως έχει φέρει τεράστιες προκλήσεις και μεγάλες ανισότητες μεταξύ χωρών και εντός των χωρών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη θα κατανέμονται επαρκώς μεταξύ ανθρώπων και χωρών. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα βασίζεται σε κανόνες και δεν θα εφαρμόζει αποκλεισμού. Θα πρέπει να είναι ένα ε, όχημα αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασία, ε, την εκρίζωση τη φτώχεια και των ανισοτήτων. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλε τι ανάγκε ε, τη ισότητα τη παγκοσμιοποίηση μόνο μέσω του ODI. Χρειάζονται και πρωτοβουλίε απαραίτητε για την ένταξη των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών στην παγκοσμία οικονομία. Επιπλέον, ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση του θεματολογίου 2030 διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε συνοδευτικά μέτρα και οικονομική στήριξη. Όλα αυτά πρέπει να υλοποιούνται με τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε με τις τρίτες χώρες ώστε να υποστηρίζουμε τις δικές τους προσπάθειες να τηρήσουν τα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον και για τα κοινωνικά θέματα. Πρέπει επίση να υπάρχει πλήρη διαφάνεια στι εμπορικέ συμφωνίε και πλήρη συμμετοχή των κοινωνιών, των πολιτών, των χωρών εταίρων με τι οποίε διαπραγματευόμαστε και συνάπτουμε συμφωνίε. Οι αναπτυσσόμενε χώρε, ειδικότερα οι αφρικανικέ, ακόμα βρίσκονται στο περιθώριο ε, παγκοσμίω. Πρέπει να τι υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε εκεί τη δημιουργία μιας ε, πραγματικής ενδοφρικανικής αγοράς ε, και να κάνουμε πραγματικότητα τις φιλοδοξίες ε, που έχουμε για αυτό το χώρο. Επίσης να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη της μετανάστευσης και της κινητικότητας, να υποστηρίξουμε τις αφρικανικές χώρες για να ενισχυθούν οι παραγωγικές και μεταπητικές τους δυνατότητες, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και η συμμετοχή τους στην παγκόσμια αγορά. Κάθε χρόνο τεράστια, έχουμε τεράστιες οικονομικές ροές που βγαίνουν από την Αφρική λόγω φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, ε, πολύ συχνά από τις δικές μας εταιρείε. Έτσι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν αποτελεσματικά εργαλεία καταπολέμησης της ε, φοροαποφυγής παγκοσμίω και να ενισχύσουμε τη φορολογική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες και σε θέματα εσωτερικής κινητοποίησης των πόρων. Οι δικές μας τροπολογίες θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση για το πρώτο αυτό σχέδιο. Προσβλέπω μια επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και όλους τους σκιώδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Χόιμπου. Ε, Κύριε Χόιμπου, ευχαριστώ πολύ και τον Ταν Μπρέντα για την καλή βάση που έχουμε τώρα στη γνωμοδότησή του. Και εμείς οι πράσινοι θέλουμε να ενισχύσουμε κάποια σημεία και να συμπληρώσουμε λίγο κάποια άλλα για να αλλάξουμε λίγο τις τάσεις, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε στην έκθεση. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά σημεία. Για το συντάκτη της γνωμοδότησης παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο ο ιδιωτικός τομέας στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Υπάρχει όμως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα για να αρθεί αυτή η ασυμμετρία. Γιατί οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις έχουν πάρα πολλά δικαιώματα και σχεδόν καθόλου υποχρεώσεις. Αυτό κάπως θα πρέπει να αλλάξει και να εξισορροπηθεί και να γίνεται ρητή μνήα και να παίρνει θέση και ο εισηγητής για τη σύμβαση του άρα να του συμπεριλάβει και στην έκθεσή του. Επίσης παρατηρούμε ένα κατακαιρματισμό. στον τρόπο με τον οποίο συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίες. Και χαίρομαι που τονίζει ο εισηγητής ότι χρειαζόμαστε την πολυμερή προσέγγιση. Αυτή είναι και δική μας θέση των πρασίνων και συμφωνούμε πάρα πολύ με αυτό. Έχουμε πολλές διμερείς συμφωνίες έτσι, και με αυτόν τον κατακαιρματισμό ε, αποδυναμώνουμε τον ΠΟΕ και επιδεινώνουμε την κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες αντί να τη βελτιώνουμε. Αυτές οι διμερείς λοιπόν εμπορικές συμφωνίες συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις ενώ τα πλεονεκτήματα των κανόνων του ΠΟΕ παρακάμπτονται με αυτόν τον τρόπο και ε, χαίρομαι που το τονίζει αυτό η γνωμοδότηση. Στη συνέχεια πιστεύω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως είπε και η Έλλη Σλάιν προηγουμένως, χρειάζονται περισσότερο περιθώριο γυρισμών για να αναπτύσσουν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές και να θέτουν τις δικές τους προτεραιότητες, ενδεχομένως να τις διαμορφώνουν και καλύτερα. Παράδειγμα, οι δυνατότητες παραγωγής στη γεωργία ή στην τοπική γεωργία μπορούν να ενισχύονται όταν το αποφασίζουν αυτό. Να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμών για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι κανόνες του ΠΟΕ προβλέπουν έκτακτες και ε, προτιμησιακές ρυθμίσεις για τα αναπτυσσόμενα κράτη. Ε, η μεταφορά στη πράξη όμως χωλαίνει και θα πρέπει να βελτιωθεί για να έχουν, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερες δυνατότητες να παίρνουν αποφάσει και να ε, αναπτύσσονται και να διαφοροποιούν την οικονομία του στα αναπτυσσόμενα κράτη. Και προ την κατεύθυνση αυτή θα κάνουμε και τροπολογίες. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δύο λόγια, το κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην γνωμοδότηση και ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. σε εμπορικέ συμφωνίε έχει την πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει και ρήτρε για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντίστοιχα κεφάλαια. Και χαίρομαι που όλα αυτά είναι και δεσμευτικά πλέον. Αντίστοιχη όμως προσπάθεια πρέπει να γίνει για την παρακολούθηση όλων αυτών και όταν δεν τηρούνται να ε, υπάρχουν και κυρώσεις που να επιβάλλονται. Επιστημιστική ασφάλεια, επίσης, είναι ένα ιδιαίτερα προσφυλές μου θέμα. Οι τιμές και οι αγορές είναι ρευστές. Και έχουμε και νέα διάνοιξη των αγορών. Αυτό μπορεί να ε, συνιστά απειλή ε, και κίνδυνο για την επιστημιστική ασφάλεια και τις αγορές ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τώρα δεν θα έχουμε ε, συμφωνίες ε, εταιρικέ σχέσεις όπως είναι η EPA. Ε, χρειάζεται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση όλων αυτών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει και την αναπτυξιακή της πολιτική θα πρέπει να δείξει συνέπεια με και αλληλεγγύη με τις χώρες του Νότου, έτσι ώστε ε, να μπορούν να διαφοροποιούν την παραγωγή τροφίμων οι χώρες αυτές και να προστατεύουν και κάποιους κλάδους της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί και αυτό στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και πάλι τον συντάκτη και όπως είπαμε θα υποβάλουμε αντίστοιχε τροπολογίες από την πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση ΤΕΠΚΟ. Θέλετε κάτι να πείτε εδώ, να προσθέσετε. Αξέλ Πουζά. Ζουλικά. Καλησπέρα. Γιούλικα πίσω. Trade σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και την επικοδομητική γνωμοδότηση η οποία τονίζει το θετικό αντίκτυπο των συμφωνιών για την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν μιλούμε για συνοδευτικά μέτρα στις ε, συμφωνίες και την ανάπτυξη των, ε, της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη και την, το συνδυασμό της ε, αναπτυξιακής βοήθειας έναντι εμπορίου που δίνεται και των λοιπόν προγραμμάτων υποστήριξης Αξέλα de από την ΤΕΦΚΟ. Θα ήθελα απλώ να τονίσω αυτά που είπε η συνάδελφος. Έχουμε μια νέα ανακοίνωση της Επιτροπής Ενίσχυση Έναντι Εμπορίου η βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια. Σας ε, την παρουσιάσαμε άλλωστε πριν από μερικού μήνε. Και αποτελεί πιστεύω ένα πολύ σημαντικό ε, έγγραφο ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση και το θέμα που έχετε εδώ. Η στόχη της είναι διτή. Αφενός με ένα συνδυάζει καλύτερα την ε, βοήθεια εναντί εμπορίου, που είναι το 1 τρίτο άλλωστε τη ε, αναπτυξιακή βοήθεια συνολικά. Και εδώ έχουμε συμφωνίε ε, και βέβαια τη ΣΥΠΑ, αλλά και τη Συμφωνία ε, των Προτιμήσεων και του τους στόχου, και στόχο έχει να ενισχύσει το παραγωγικό δυναμικό των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών ώστε να μπορούν να υποφελούνται από τις εμπορικές προτιμήσεις όταν τους χορηγούνται και όπως τους χορηγούνται. Βέβαια, αν δεν έχουν προϊόντα για διάθεση του εμπόριο, δεν μπορούν να υποφεληθούν από τις εμπορικές προτιμήσεις. Αυτό είναι το πνεύμα λοιπόν της ανακοίνωσης, με μια επικαιροποιημένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά όχι μόνο την Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη. στο θέμα της θεθάσευσης της ε, παγκοσμιοποίησης, της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ κρατών αλλά και στο ιστορικό αυτών. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο με την ε, πολιτική αυτή και ήθελα να το τονίσω ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε, Μπογκτάν; Όχι, απλά ότι ο κύριο εισηγητή θα τα λάβει όλα υπόψη, όπω λέει και στο κείμενό του. Έχουμε κάποια περιπτώσει όπου δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε όλε τι ιδέε στην έκθεση αυτή, αλλά θα λάβουμε υπόψη στο βαθμό του δυνατό όλε τι προτάσει και συστάσει όλων των σκιωδών. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία είναι η Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 11 θα ψηφίσουμε τον Αύγουστο μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, έχουμε κάποιους προσκεκλημένους. Ε, εδώ θα καλέσω τους ε, προσκεκλημένους μας εδώ στο επόμενο σημείο για το Grand Bargain. Επίσης μας έχουν δώσει ένα φίλο ενημερωτικό οι, οι διερμηνείς ε, με κάποιες πληροφορίες για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε με τη διοίκηση. Θα πρέπει να το έχετε λάβει. Καθώ έρχονται εδώ οι προσκεκλημένοι, Ερικέ, να πω ότι από την ε, Γενική Διευθύνση ΕΚΟ στι ανακοινώσει ε, μάθαμε ότι η Κομισιόν τώρα δημοσίευσε την έτσι ανακοίνωση για την εκπαίδευση και τι περιοχέ έκτακτη ανάγκη, τι καταστάσεις έκτακτη ανάγκη. Είναι η πρώτη φορά που ε, κυκλοφορεί αυτή η πολιτική. Εδώ και χρόνια μας απασχολεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Πάμε στο σημείο 7 αφορά τα αποτελέσματα της δεύτερης ετήσιας συνάντηση των συμβαλωμαρών στη Συμφωνία Grand Bargain που συνήθη κατά την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη κορυφή του 2016. Συμφωνία που συνάφθη στο πλαίσιο της 26ης Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής μεταξύ των 18 μεγαλύτερων χορηγών και 48 ε, παρόχων ε, με στόχο να παρέχεται μεγαλύτερη βοήθεια στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Μετά από την υπογραφή προσθέθηκαν και άλλοι υπογράφοντες. Όταν εγώ διάβασα τον όρο Grand Bargain, μεγάλο στοίχημα, φαινόταν κάπως περίεργο για ένα εργαλείο ανθρωπιστικής βοήθειας. Και δεν κατάλαβα πολύ ακριβώς τι εννοούσαν. Grand Bargain στα αγγλικά σημαίνει και ε, κάτι που βρίσκει κανείς σε ευκαιρία, σε ένα μαγαζί, σε καλή τιμή. Εξηγήστε μας λοιπόν εδώ τα βασικά. Τι είναι το ground bargain, ε, η μεγάλη αυτή ευκαιρία, τι... Ε, σε τι μας βοηθάει. Έχουμε εδώ τους ε, εκπροσώπους της Κομισιόν που θα μας δώσουν τις απόψεις τους, ο Ερίκε Τράουτμαν και η Μαγκαλή Μουλόγκ ε, να μας εξηγήσουν ακριβώς τι είναι το grand bargain και τι σημαίνει σε, πρακτικού, σε απλά λόγια και στην πρακτική. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα στους συναδέλφους και ε, στην Πρόεδρο. Ήρθατε εδώ να σας εξηγήσουμε το grand bargain. Ναι, δεν ήταν Άγγλος αυτός που το επινόησε, γι' αυτό ίσως είναι λίγο περίεργη λέξη. Να σας παρουσιάσω λίγο α, τις βασικές πληροφορίες. Το grand bargain είναι ένα από τα τρία μέρη του υψηλού επίπεδου πανέλ για τη χρηματοδότηση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2016 πριν από την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφή. Διερευνούσε τρόπους βελτίωσης της χρηματοδότησης για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το ένα ονομάστηκε συρρήκνωση των αναγκών Ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα χρειάζονταν λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο. Δυστυχώς αυτό έχει αποτύχει, όπως είναι σαφές, και ουσιαστικά έχουμε περισσότερη ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά τουλάχιστον ε, ήταν ε, ένα κομμάτι της σχετικής έκθεσης. Το άλλο ονομαζόταν διευρύνοντας τη βάση για την εξέβρεση χρημάτων πέραν της ε, κλασικής θεσμικής χρηματοδότησης των κλασικών δωρητών Ούτε αυτό πάει πολύ καλά. Πέρυσι για πρώτη φορά η χρηματοδότηση ε, αυτή ε, μειώθηκε οπότε επιστρέφουμε στα κλασικά, στους κλασικούς χορηγούς ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδούς, Αμερικανούς είχαμε και κάποιο άνοιγμα από τους Άραβες αλλά αυτό έχει κινητοποιηθεί λίγο τώρα απομένουν πολλά φυσικά να γίνουν γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να συμμετέχουν και ιδιώτες οι ο τομέα των ασφαλίσεων, ειδικότερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση ετοιμότητα. Όλες, όλα αυτά τρέχουν αυτή τη στιγμή και μετά το τρίτο κομμάτι ήταν το Grand Bargain όπως αναφέρθηκε που εξέταζε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας και πώς μπορούσε να βελτιωθεί ουσιαστικά για να απλουστευθούν περισσότερο οι διαδικασίες. Το Grand Bargain ε, επινοήθηκε ε, για να χαρακτηρίσει 10 διαφορετικέ ε, ροέ ε, εργασιών, στο πλαίσιο των οποίων είχαμε 51 δεσμεύσει. Εκεί υπήρξαν διάφορε διαδικασίε. Θα επανέλθουμε σε αυτό και θα σα παρουσιάσω και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε μετά από την υπογραφή του Grand Bargain στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφή στο Μάιο του 2016. Αρχικά υπογράφηκε από 32 μέρη, χορηγοί, μεγάλοι οργανισμοί του ΟΗΕ, κάποια δίκτυα ΜΚΟ. Τώρα έχουμε 59 υπογράφοντες, περιλαμβάνουν πολλές ε, επιμέρους ε, ΜΚΟ αλλά και οργανισμούς όπως το ε, Enia Network που εκπροσωπεί τοπικούς οργανισμούς του Global South όπως το ονομάζουμε που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Κατά βάση αυτό που έχει συμβεί και αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα είχαμε την ετήσια συνάντηση ε, του Grand Bargain και πριν ε, από την ετήσια συνάντηση έγιναν αυτοαξιολογήσεις ε, σε σχετικές εκθέσεις από τα μέρη. Πώς θεωρούν ότι ελοπίσαν δηλαδή τις δεσμεύσεις επιπλέον. Έχουμε ένα θέση και μια ανεξάρτητη ετήσια έκθεση για τον Grand Bargain. Κάτι πολύ επαναστατικό θεωρούμε, διότι ουσιαστικά ζητάμε από κάποιους, κάποιον εξωτερικό οργανισμό να αξιολογήσει την πρόοδό μα. Δεν υπάρχει τέτοια εγχείρημα σε κανέναν ε, διεθνή οργανισμό. Ήταν πολύ χρήσιμο. Εδώ μπορείτε να βρείτε την ετήσια έκθεση για τη φετινή χρονιά. μόλι δημοσιεύτηκε από το Overseas Development ε, Institute και το Humanitarian Policy Group. Πολύ καλή δουλειά έχει γίνει εδώ και σα δίνει μια καλή εικόνα του που βρισκόμαστε. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Υπάρχει καλή πρόοδος ε, ε, σε κάποιες δευτερεύουσες ε, ροές εργασίας. Αλλού απομένουν να γίνουν πολλά. Γενικά, όπως βλέπουμε, έχουμε μεγάλη πρόοδο στα συστήματα μετρητών. Ουσιαστικά και η DJ προωθεί όλο και περισσότερο αυτά τα συστήματα cash, τα συστήματα μετρητών και έτσι παρέχουμε ενημέρωση στα κράτη-μέλη και σε διάφορα μέρη για το πώς αυτό γίνεται. Ξέρετε, έχουμε το σχετικό δίκτυο στην Τουρκία για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ιορδανία, στο Λίβανο και εκεί αυτή η βοήθεια σε μετρητά είναι ο βασικός τρόπος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2017 η DJECO δαπάνησε 35% του συνολικού προπολογισμού ε, στην περιοχή ε, Μένας, ε, βοήθεια σε μετρητά. Επίσης έχουμε βελτίωση σε θέματα διαφάνειας 100% της επιτόπου χρηματοδότησης στην βάση δεδομένων γιατί και στους συνολικούς δείκτες αναφέρεται έως και 70% σε, όλα τα, σε όλους τους τομείς του Grand Bargain υπάρχει όλο και περισσότερη πολυετής χρηματοδότηση μας ζητούσαν πολυετής, πολυετής χρηματοδοτήσεις και από τη Σύνοδο δεν μπορούσαμε να ανανεώνουμε τις συμβάσεις κάθε χρόνο οπότε ο στόχος για την Κομισιόν είναι 15 20% πολυετής συμβάσεις το 2018 και προσπαθούμε να το ενισχύσουμε, αλλά υπάρχουν και πιο γενικά θέματα πολιτικής όπως η σύνδεση μεταξύ ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Ε, μεγάλη ροή και αυτή για τον Grand Bargain, γίνονται πολλά εκεί. Κράτη μέλη θα γνωρίζουν διάφορα πιλωτικά έργα που έχουν συζητηθεί, κάποια ειδικά workshop που ε, αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκή Ένωση, γραφεία της ΕΚΟ και εκπρόσωποι σε διάφορες χώρες πιλωτικές έχουν οργανώσει. Γίνονται πολλά δηλαδή εκεί. Πιο δύσκολο είναι η τοπική προσαρμογή, το localization, αυτός ο στόχος του Grand Bargain υπολογίζει ότι το 20-25% της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης παγκοσμίω θα πρέπει να υλοποιείται από τοπικούς φορείς, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι χορηγοί ε, απέχουν αρκετά από αυτό. Στη δική μα περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι η νομική βάση τη ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μα επιτρέπει να χρηματοδοτούμε άμεσα ε, φορεί που δεν έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε αυξήσει του φορεί ε, που λαμβάνουν χρηματοδότηση από έναν διάβλο μόνο μέσω μια αντί για να τη λαμβάνω από δύο-τρει διαφορετικέ πηγέ. Έχουν γίνει πολλέ βελτιώσει δηλαδή, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν. Η Κομισιόν έχει χρηματοδοτήσει διάφορε ασκήσει ε, ανάπτυξη ικανοτήτων με τοπικού φορεί. Του βοηθά να υλοποιήσουν και ειδικέ ε, στρατηγικέ ε, χρηματοδότηση που μπορούν να ξαναχρησιμοποιήσουν οι δωρητέ στο μέλλον. Και η τελευταία ροή εργασιών είναι η αξιολόγηση αναγκών. Πολύ δύσκολη διότι γίνονται πολλά καλά πράγματα σε τεχνικό επίπεδο, ενώ σε πολιτικό επίπεδο τα πράγματα παραμένουν δυσχερή. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ακόμα σε μια κατάσταση όπου κάθε ανθρωπιστικός οργανισμός, ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ο Ερυθρός Σταυρός, ο καθένας κάνει τη δική του αξιολόγηση της κρίσης και ε, τη δική του στρατηγική ε, Χρηματοδότηση ε, ανθρωπιστική ε, και ζητά το δικό του κομμάτι τη πίτα από του δωρητέ, οι οποίοι έχουν πρόβλημα διότι δεν μπορούν να αποφασίσουν πώ θα κατανέμουν αυτά τα κονδύλια και επιπλέον λαμβάνουν αιτήματα από τι πλευρές και προσπαθούν να εξορροπήσουν μεταξύ τη κρίση Συρία, την Τουρκία, τη Ρογίνγκα, τι χώρε της Αφρικής. Τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά πολύπλοκα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για το πού θα εστιάζουμε ή πώ θα καταναμούμε ισότιμα τα χρήματα. Οπότε αυτή η ροή εργασιών ίση αξιολόγηση θα μα βοηθήσει να καθορίζουμε πιο σωστά τι προτεραιότητε σε ολόκληρο το σύστημα, ώστε να χρηματοδοτούμε βάσει των προτεραιοτήτων. Και όπω είπατε, Λίντα, αυτό θα μπορούσε να αφορά την εκπαίδευση σε χώρε που αντιμετωπίζουν εκτακτή ανάγκη κτλ. Είναι δύσκολη αυτή η εξισορρόπηση Καθώ πλησιάζω προ το τέλο τη παρουσίασή μου κάποιε αξιολογήσει που έχουμε κάνει για τι διαδικασίε στην συνάντηση στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα αντιληφθήκαμε ότι εξακολουθεί να είναι δυναμική αυτή η διαδικασία, εξακολουθεί να θεωρείται πιθανό όχημα αλλαγή και βλέπουμε ότι έχει γίνει, έχουν γίνει πολλέ αλλαγέ ε, με το Grand Bargain και ορισμένε διαδικασίε ε, και οι διαδικασίε ε, υποβολή εκθέσεων μα βοηθούν να μην ξεχνάμε αυτά τα θέματα. Ωστόσο, παρατηρούμε κάποιε δυσκολίε όσον αφορά την αποτίμηση αυτών των ε, κερδών από την αποτελεσματικότητα, διότι και οι οργανισμοί και εμείς δυσκολευόμαστε να πούμε ότι αν περάσουμε ας πούμε από έναν τύπο χρηματοδότηση σε cash, σε μετρητά, πόσα εξοικονομούμε και πόσο πιο αποτελεσματικά δράμε. Οπότε έχουν ακόμα πολλά να γίνουν σε θέματα δικτών, ε, και το αφήγημα το πώς παρουσιάζουμε όλο αυτό στον Ευρωπαίο Φορολογούμενο είναι ένα θέμα για το πώς παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για το πώς έχουμε βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε τώρα. Ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα για την Κομισιόν είναι ότι αν κάνουμε ε, πιο ευέλικτη τη χρηματοδότηση των μεγάλων οργανισμών ε, των εθνών Θέλουμε να κινηθεί και προς τα κάτω αυτή η ευελιξία. Δεν έχει νόημα η ΕΚΟ να αφιερώνει σε ειδικό σκοπό συγκεκριμένα κονδύλια εάν μετά ο ΙΕ τα δεσμεύει για διεθνείς ΜΚΟ και μετά για τοπικές ε, ΜΚΟ δεν, δεν κερδίζουμε τίποτα σε θέματα αποδοτικότητας του σύστημα οπότε εξακολουθούμε να το εξετάζουμε όσον αφορά στους συνολικούς ε, δείκτες πρόξη που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για την μέτρηση της ε, ε, αποτελεσματικότητας. Τώρα χρησιμοποιούμε το λόγο το πόσο χρήματα λαμβάνει ο δικαιούχος επιτόπου. Αυτό το είχαμε ξεκινήσει με το ESSN και την Τουρκία και την ιδέα ότι όσο περισσότερα χρήματα λαμβάνει ο δικαιούχος τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Όσο δηλαδή λιγότερα γενικά έξοδα διοικητικά έχουμε, τόσο πιο επιτυχή θεωρούμε τη διαδικασία της χρηματοδότησης και τώρα έχουμε λόγους ε, στην Τουρκία επίπεδου 85-15, 90-10, τέτοιους λόγους. Ε, οπότε θεωρείται αρκετά επιτυχής εκεί η διαδικασία. Τα επόμενα βήματα. Η συνάντηση την περασμένη εβδομάδα κατέληξε σε κάποιους στόχους για την ε, διαχειριστική ομάδα που οργανώνει τις εργασίες και το eminent person που είπαμε, το, η εξέχουσα προσωπικότητα, η Κριστέλνα Γεωργίευα, όπως ε, διορίστηκε, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι ροές εργασιών, να, απλο, να απλουστευτούν και διάφορες δεσμεύσεις επίσης και να ασκηθεί και πίεση σε πολιτικό επίπεδο, ώστε η διαδικασία αυτή να προβληθεί επαρκώς, ώστε να δείξουμε στους διάφορους ενδιαφερομένους ότι υπάρχουν και περαιτέρω κέρδη πέραν των λόγων. Κάποια στιγμή σαφώς θα πρέπει να δούμε και σαφή αποτελέσματα, τα αποτελέσματα ε, ότι έχουν επιτευχθεί δηλαδή οι δεσμεύσεις του Grand Bargain από πλευράς Κομισιόν. Ε, προφανώς θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και όλες αυτές τις πληροφορίες τις συζητήσεις ε, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την αναθεώρηση της DJ αναθεώρηση των σχέσεών της με τους εταίρους της που ξεκινούν τώρα. Και θα πάρουμε δηλαδή όλα αυτά τα μαθήματα από το Grand Bargain και θα τα χρησιμοποιήσουμε για τις επόμενες συζητήσεις. Δίνω το λόγο στη Μαγκαλή. Ευχαριστώ πολύ. Μαγκαλή Μογλό. Όπως είπαμε από την ε, ΜΚΟ Voice που εκπροσωπεί τους ε, εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκερέρο Σαλόμ ε, για την πρόσκληση και για τη συνεισφορά του. Πριν περάσω στη συμφωνία Grand Barking, για όσοι δεν μας γνωρίζετε το Voice, είμαστε ε, ένα δίκτυο ανθρωπιστικών ΜΚΟ που ε, έχουμε έδρα την Ευρώπη, 86 οργανώσεις. περισσότερες αν όχι όλες είναι εταίροι και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Δράσης, ΕΚΟ. Όπως ακούσαμε είναι 51 δεσμεύσεις το Grand Bargain, αυτή η μεγάλη συμφωνία είναι πολύ καινοτόμα. Συνεργάζονται οι μεγάλοι ε, ανθρωπιστικοί οργανισμοί σε ίσους όρους 51 στόχους έχουμε σε 10 διαφορετικά θέματα και από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών οργανώσεων, εμείς πώς το βλέπουμε, ότι οι δωρητές δεσμεύονται να δώσουν πολλά χρήματα ε, κάνουν ωραίες υποσχέσεις, τα προσημειώνουν και από την άλλη όμως έχουμε τους ε, οργανισμούς που τα υλοποιούν όλα αυτά, που είναι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δεσμεύονται να είναι πιο αποτελεσματικοί, να ε, βελτιώσουμε ε, τη δράση μας και συλλογικά να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα χρήματα και μετρητά για να συμμετέχουν περισσότερο οι τοπικοί εταίροι και να υπάρχει γενικότερα μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη υλοποίηση και συμμετοχή των δικαιούχων από την αρχή στο σχεδιασμό. Overall, what's the, the NGO's perspective on the ground ε, πώς το βλέπουν λοιπόν αυτό το μεγάλο στίχημα η Μίκιο. Ε, γενικά θετικά, γιατί είναι μοναδική αυτή η προεπτική και είναι και μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που εδώ και καιρό έχουμε εντοπίσει στο σύστημα και είναι πολύ καινοτόμια αυτή η προσπάθεια, αλλά και με τρόπο πολύ πιο μετρήσιμο. Δεσμεύονται ε, τα συμβαλόμενα μέρη όσοι έχουν υπογράψει τη συμφωνία σε αιτήσια βάση να κάνουν εκθέσεις και αναφορές. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο ε, ακριβώς για να λογοδοτούν κιόλας κατά πόσο έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν είναι πολύ σημαντικό. Συμμετείχαν σε μια διαβούλευση την τελευταία διετία η ΜΚΟ για να καταλήξουμε εκεί. Είναι πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες, υπερβολικά πολλές και αυτό είναι μειονέκτημα γιατί οι ΜΚΟ έχουν περιορισμένους πόρους και ε, δυναμικό ανθρώπινο και οικονομικούς πόρους και χρόνο λίγο και βλέπουμε ότι στην ίδια θεματική ενότητα δεν γίνεται μεγάλη πρόοδος και καμιά φορά έχουμε αντιπαραγωγική παρουσία και ε, εμπόδια. Επίσης, γενικότερα, η συνεργασία μέχρι τώρα ε, θεωρείται ότι ήταν μια κλειστή λέσχη μεταξύ κάποιων ε, συγκεκριμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων και πολλές μικρές οργανώσεις δεν είχαν πρόσβαση και πολλές φορές οι ντόπιοι δεν είχαν πρόσβαση. Και είχαν την αίσθηση ότι ήταν ε, ε, παραγωνισμένοι. Και είναι καλό λοιπόν που το δίκτυο αυτό των μη κυβερνητικών οργανώσεων συμμετέχει σε αυτή τη ε, μεγάλη συμφωνία και το μεγάλο στοίχημα Grand Bargain. Τι λέει λοιπόν το δίκτυό μας Voice. Συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια Grand Bargain από την αρχή. Είναι ε, τα αποτελέσματα της συνεργασίας στο πάνελ υψηλού επίπεδου για ε, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη χρηματοδότηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει τέτοια μεγάλη προσήλωση και δέσμευση σε αυτή την προσπάθεια και ενθουσιασμός να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και να αυξηθούν και οι δωρητές. Ως δίκτυο εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα μέλη μας. Ε, να αρχίζει μια συζήτηση για να κατανοούμε ποια είναι η επιχειρησιακή ε, πραγματικότητα και αυτά να μεταφέρονται στη συζήτηση για τη χάραξη πολιτικής. Να γεβαιρωθεί αυτό το χάσμα και να προωθηθούν και διάφορες ε, πρωτοβουλίες στον ε, ΜΚΟ, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, συνεργαζόμαστε με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλα δίκτυα και οργανισμούς έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη θέση των ΜΚΟ παγκοσμίω. Και πρόσφατα, πριν την ετήσια έκθεση, δημοσιεύσαμε ε, μαζί με ένα άλλο δίκτυο που εδρεύει στη Γενέβη μια κοινή θέση μας, μια ετήσια συνάντηση. Ε, είχαμε και κοινή δήλωση όλων των δικτύων ΜΚΟ. έχουμε μια task force όπου συμμετέχουν 47 ΜΚΟ που συνεργάζονται με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ και έξι μήνες συζητούμε για το σχέδιο Grand Parking. Σε 10 θεματικές ενότητες, όπως είπαμε. Η χρηματοδότηση έχει τώρα όρους και προϋποθέσεις. Και ακριβώς επειδή ε, τώρα συνεχίζουμε μια δουλειά που έχουμε κάνει στο παρελθόν, όχι μόνο για την απλούστευση, που είμαστε ακρεφνώς υπέρ ε, της απλούστευσης για λόγους ε, αποτελεσματικότητας, θέλουμε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χάρη στην εφαρμογή ε, κοινών ε, στόχων αναφοράς και υποβολής εκθέσεων, που είναι μία από τις δεσμεύσεις στο Grand Bargain και θέλουμε καλύτερο σχεδιασμό και καλύτερη χρηματοδότηση είναι από τις μεγάλες μας προτεραιότητες. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή με πρόσβαση στην ενημέρωση, με πληροφορία και πρόσφατα λανσάραμε και μια σχετική στο σελίδα την περασμένη εβδομάδα στην ετήσια έκθεση και θα διοργανώσουμε και μια σειρά από εργαστήρια για να δούμε οι φορείς που οι συνεργάτες μας τόπου πώς απαντούν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν δύο χρόνια μετά και στη Νέα Υόρκη και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις καταλήγουμε ότι είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για τη συμφωνία Grand Parking. Και ευχαριστώ τον Ενρίκη Γκερέρο που βοήθησε πάρα πολύ. Βεβαίω υπήρχαν αυτέ οι συμφωνίε για τη συμμετοχή, αλλά τώρα έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα το θέμα των μετρητών, το θέμα τη διάσταση του φύλου, το θέμα τη συμμετοχή στον ΜΚΟ που υπογράφουν τη Συμφωνία Grand Bargain και αυτό είναι απόδειξη. Έχουμε σαφή προγράμματα δράσης και προσπαθούμε να μεταφράσουμε τις δεσμεύσεις μας σε συγκεκριμένη δράση που πρέπει να αναλυφθεί ε, το επόμενο διάστημα. Τώρα μπαίνουμε σε μια φάση εφαρμογής αυτή τη χρονιά. Δεν θέλουμε η συμφωνία Grand Bargain να ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα, γιατί χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοθούν οι διαδικασίες. Και δεν είναι και πολλά τα κονδύλια που έχουν προσημειωθεί για την επένδυση εκεί. Όλα αυτά είναι δαπανηρά ε, η διαφάνεια έχει ένα κόστος για να προσαρμοστούν τα εσωτερικά συστήματα μιας μη κυβερνητική οργάνωσης στα διεθνή στάνταρ και τις προδιαγραφές. Δεν χρειάζεται, ε, δεν φτάνει ένας χρόνος μάλλον, χρειάζεται περισσότερο διάστημα. Ε, λοιπόν, οι δεσμεύσει αυτέ θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα, χειροπιαστή και θα πρέπει όλοι οι υπογράφοντε τη συμφωνία αυτής να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, την πολυμερή και με πολλούς ενδιαφερόμενους. Και στην πράξη, είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε στην πράξη πώς θα μεταφραστούν όλα αυτά και πώς θα συνδυαστεί το Grand Bargain με ε, τις διάφορες πρωτοβουλίες δωρητών ε, αποδεκτών βοήθειας. Ε, ξέρουμε και τον Nexus όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς το βλέπουμε εμείς από το δικτύο Voice και πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση και γίνονται συζητήσεις για τη μελλοντική χρηματοδότηση των ΜΚΟ από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Είναι μοναδική ε, η ευκαιρία, η αναθεώρηση ε, του χρηματοδοτικού προγράμματος για να ε, δούμε πώς γίνονται οι εκθέσεις, πώς γίνεται η πολιτική χρηματοδότηση, πώς οργανώνεται και πώς υποστηρίζεται το σύστημα. Εκεί μας βοηθούν οι αξιολογήσεις της Γενικής Διεύθυνσης έχω και συστάσεις της δικής σας Επιτροπής, αλλά και χάρη στο δημοσιονομικό κανονισμό, το πρόσφατο που ενέκρινε ή που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, that you can see. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα τα βρείτε και στο δημοσιονομικό κανονισμό και στο Grand Bargain. Και είναι καλό και σημαντικό να υπάρχουν αυτά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εταίρων, το λογιστικό έλεγχο των δικαιούχων. Υπάρχει και πολύ μεγάλος χώρος για απλοποίηση των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των ε, εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δηλαδή γιατί είναι και η κατάσταση διαφορετική από ε, χώρα σε χώρα και από δράση σε δράση. Ποιος ε, είναι ο ρόλος που θα μπορούσατε εσείς να παίξετε η Επιτροπή σας στο επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, να παρακολουθείτε ε, την επίπτωση του δημοσιονομικού κανονισμού και στην εφαρμογή του. Για ΜΚΟ, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι και μια κρίσιμη ε, ευκαιρία να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα ε, του αυξανόμενου χάσματος η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν είναι μόνο αυτή η συμφωνία Grand Parking, αλλά είναι και ε, το πάνελ υψηλού επίπεδου που έχει κάνει κάποιες συστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί ο προπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Κάθε χρόνο η Επιτροπή σας, ΔΕΒΕ, είναι πάρα πολύ δραστήρια στις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό και υποστηρίζεται ε, τις αιτήσει μα για χρηματοδότηση και για τις πληρωμέ και για την ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτό είναι εκ των όνου για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και υπάρχει και το παγκόσμιο, η Παγκόσμια Σύνοδος για την ανθρωπιστική βοήθεια. Καλή αποδοτικότητα, καλή αποτελεσματικότητα, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να λησμονούμε ε, ε, τι αιτίε των ανθρωπιστικών κρίσεων. Καλέ είναι οι συζητήσεις αυτές που γίνονται για την ε, υλοποίηση των δεσμεύσεων στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφή, ε, ε, θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι η τελευταία σας παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου, ε, δεδομένου και του χρονισμού Μιλήσαμε για διαχείριση, μιλάμε για προγράμματα, αλλά βέβαια έχουμε τα κύρια πολιτικά ζητήματα που τραβούν τον ενδιαφέρον του τύπου και είναι οι μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων που από τα σπίτια τους φεύγουν για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από τη φτώχεια, από την κατάρρευση των κρατικών δομών. Αυτό και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα και είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος με τον οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες κυβερνήσεις. Μας είδαμε από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής εχθές εδώ στις Βρυξέλλες που μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Θα μας πείτε ίσω αργότερα θα μάθουμε περισσότερα. Ε, είδαμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, τι συνέβαινε όταν χωρίζαν τα παιδιά από του γονεί του. Κεντρική Αμερική εκεί για άλλα, με άλλα θέματα και προβλήματα. Ε, γίνεται λόγος για τη Βενεζουέλα νωρίτερα. Φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του λοιπόν. Επομένω έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία και το να την ε, υλοποιήσουμε, να την αντιμετωπίσουμε με τρόπο επιτυχημένο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ενρίκε Χερέρο όμω, που είναι ο εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Τράουτμαν. ελά, και την ε, άλλη ομιλήτρια για, για την ενημέρωση. Γιατί το λένε Grand Bargain, για είναι σαν Great Britain. GB για κάποιον άλλο λόγο. Δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Σοβαρά όμως τώρα γνωρίζω τη Voice που είναι ένα ε, καταπληκτικό δίκτυο και πρωταγωνιστικό στην ανθρωπιστική δράση. Και βλέπουμε πώς αξιολογεί την εφαρμογή του Grand Bargain. Το Κοινοβούλιο έστειλε την προσωπία στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφή στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχα κι εγώ εκεί. Και θυμίζω, ε, θυμάμαι μάλλον την ε, στιγμή που έγινε η παρουσίαση του Grand Bargain με χώρες που αναλάμβαναν επιπλέον δεσμεύσεις, πέραν των ε, δεσμεύσεων που είχαν ήδη αναλάβει και που θα μπορούσαν από κοινού όλες οι χώρες να υλοποιήσουν, των Ηνωμένων Εθνών δηλαδή. Και αν θυμάμαι καλά, οι δύο βασικοί στόχοι ήταν πρώτον, να καταλήγουμε σε ε, συμφωνίες αποτελεσματικές και έτσι, λειτουργικές, γιατί είναι δύσκολο να συμφωνήσουν 179 χώρες από να συμφωνήσουν 22, για να πω τυχαία τα νούμερα. Ε, το δεύτερο πιο σημαντικό είναι πώς να προσελκύσεις νέους δωρητές. Ιδιαίτερα τις χώρες του Περσικού κόλπου και ορισμένες χώρες που εγκατέλειπαν την ε, ιδιότητα του λιγότερο ανεπτυγμένου κράτους και έμπαιναν ε, αναπτυγμένα. Και όταν οι ανθρωπιστικές κρίσεις ήταν πιο έντονες, Ε, είχαμε περισσότερες προκλήσεις, γιατί όλες οι συμφωνίες ε, είχαν σχέση με την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο χρόνια αργότερα, λοιπόν, όχι για λόγο ε, του grand bargaining, αλλά επειδή έτσι εξελίχθηκε ο κόσμος, οι ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εξίσου μεγάλες, για να μην πω μεγαλύτερες. Παρόλα αυτά όμως, η χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες δεν αυξήθηκε ουσιαστικά και σημαντικά. Και τώρα υπάρχουν χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε που μειώνουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια γενικά για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων και επίσης έχουμε και θα δούμε αργότερα σε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την περίπτωση της Λωρίδας της Γάζας, του κέρατος της Αφρικής και αλλού. Δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για να εγγυηθούμε την επιβίωση σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Τι εννοώ λοιπόν. Είναι καλή είδηση το γεγονός ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις αξιολογούν θετικά την έκβαση αυτής της διετίας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι αξιολογεί επίσης ε, στη Νέα Υόρκη θετικά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας τώρα προς τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πραγματικότητα των ανθρωπιστικών κρίσεων και προβλημάτων. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, θα πρέπει να περάσουμε από την θεσμική ικανοποίηση ε, στην ε, αντιμετώπιση, την αποτελεσματική όμως, αυτών των ανθρωπιστικών κρίσεων. Να κάνω μερικά μικρά σχόλια. Και μετά Έχω και μια μικρή παγίδα έτσι για την κυρία Τράουτμαν, ε, φιλικά πάντα, λίγο προβοκατόρικη. Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να εντάξει το Grand Bargain στις ε, επόμενες πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας θα είναι ξεχωριστό και θα μπορούμε να αγωνιστούμε και να πιέσουμε για το ίδιο αυτό το μέσο χωρίς να είμαστε σε ε, ανταγωνισμό με κάποιον άλλον στο κοινοβούλιο, με άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό σίγουρα θα είναι πιο περίπλοκο στην αναπτυξιακή πολιτική την ίδια. Και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δρομολογηθούν τα διάφορα μέσα, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα έκανε και θα χαιρόμασταν όλοι πάρα πολύ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τη στιγμή που θα αρχίσει η ειδική διαπραγμάτευση να μας βοηθήσει να δούμε ποια είναι ακριβώς αυτά τα προγράμματα οι στόχοι ή οι προκλήσεις που ε, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας με μεγαλύτερη ένταση. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αν δεν απατώμε, Δανία, Βέλγιο, Σλοβενία, που απαιτούν από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται να έχουν διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Και αν κατάλαβα καλά την κυρία Τράουτμαν, και είναι και αυτό καλή είδηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να τους βοηθήσει για να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται επιτόπου ε, τις βοήθειες και την ενίσχυση. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πρέπει να ε, εργαστούμε περισσότερο, να συνεργαζόμαστε για την εκτίμηση των αναγκών. Στις ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούμε να ανταποκρινόμαστε πάντα αντιδρώντας όταν ξεσπάνε διάφορες ανθρωπιστικές κρίσεις είναι γεγονό ότι σε πολλέ περιπτώσει και δυστυχώ είναι δύσκολο να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Όταν πρόκειται για μια θεομηνία, α πούμε. Είναι ακόμα δύσκολο να προβλέψει κανεί πώ θα εξελιχθούν οι πολιτικέ σειράξει. Αλλά ακριβώ τώρα που αρχίζουμε να συζητάμε μια επταετή αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια εκτίμηση των οικονομικών, θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή διάγνωση ε, των αναγκών, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο ως συμμετέχοντες στη μεγάλη αυτή συμφωνία στο Grand Bargain, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω λοιπόν την εξής ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κωνσταντινούπολη, όπως και όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, ανέλαβε ειδικέ υποχρεώσεις και δεσμεύτηκε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καμιά φορά Μάλλον έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει όχι απλώς ε, πώς λειτουργούν το Grand Bargain, οι άλλοι εταίροι, οι δεσμεύσεις, αλλά πώς υλοποιούνται οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κωνσταντινούπολη και τις γενικές και τις ειδικές της υποχρεώσεις ως ε, μέλος του Grand Bargain. Για τον Nexus, ε, ξέρετε ότι είναι μια αιμονή αυτή της Αναπτυξιακής Επιτροπής της δικής μας εδώ. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις είναι κρίση μακρά διαρκεία και κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντάμε με κάποια διαρθρωμένη ε, μορφή για τη βοήθεια στην ανάπτυξη. Και όχι απλώς μια επίγουσα ε, βοήθεια ανθρωπιστική πρώτης ε, ανάγκης. Καλέ είναι λοιπόν οι αξιολογήσει, οι εκτιμήσεις, πολύ δε περισσότερο όταν είναι εξωτερικές, διότι συνεισφέρουν στο να διατηρηθεί η όθηση, αυτή η ορμή που δημιουργείται τη στιγμή που αναλαμβάνουμε τις ε, αυτές οι οποίες σιγά σιγά χαλαρώνουν και χάνονται αν δεν ελέγχονται. Και τώρα η παγίδα που θέλω να στήσω στην κυρία Τράτμα. Παρακαλώ σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσετε σε αυτό που είπε το Voice. Ε, το τέλος. Τι θα κάνουμε την επόμενη διετία. Thank Ευχαριστώ. Κύριε και έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρέπει να βάλετε τα ακουστικά σας. Ο Ενρίκε ε, έκανε λόγο για μια καλή διάγνωση των αναγκών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω πρέπει να δούμε, να κάνουμε μια καλή διάγνωση και από πού θα, βρουν, θα βρεθούν τα χρήματα γιατί πολλές φορές έχουν δοθεί υποσχέσεις για κονδύλια, αλλά όταν έρθει η ώρα απλώς αλλάζουν τίτλο ή έχουν δοθεί υποσχέσεις δύο και τρεις φορές για το ίδιο ποσό, το οποίο τελικά δεν είναι διαθέσιμο. Γι' αυτό νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να διατυπώσουμε την απέτηση σαν ένα κώδικα συμπεριφοράς και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ξεκάθαρο όταν υπάρχει κρίση, όταν δεν μπορούμε να βρούμε ε, την πηγή των ε, χρημάτων, με ποιο τρόπο θα γίνει η άντληση των πόρων για να είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Ή ας μιλάμε καθαρά, ας λέμε θα δώσουμε περισσότερα χρήματα. Αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ε, δουλειά τη δική μας, τη δική σας των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρέπει ξεκάθαρα να μιλήσουμε για έναν κώδικα συμπεριφοράς και περισσότερη διαφάνεια για τους πόρους. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο το λόγο. Έχω και εγώ μια-δύο παρατηρήσεις. Ο πολιτής σχεδιασμός, πολύ σωστά είπε ο Ενρικέ, ότι χρόνια τώρα μιλούμε για την ανάγκη να έχουμε πολιετή προγραμματισμού. Και όταν επισκεπτόμαστε αυτές τις περιοχές βλέπουμε με σάρκα και το τι συμβαίνει. Είδαμε τι προγραμματισμό τι σημαίνει για την Ουγγάντα, παραδείγματι. Γιατί έχουν ένα χρόνο, έτσι. Του λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε αυτό το ποσό να δαπανίσετε και πάνε να φυτέψουν για ένα χρόνο. Φτάνει ο Μάρτιο και ο Απρίλιο. και του λένε «Α, κοιτάξτε, ε, λίγα ακόμα χρήματα μπορούμε να σα δώσουμε, αλλά πρέπει να κινηθείτε κι εσεί πιο γρήγορα». Οπότε τρέχουν, σπέβδουν να βρουν μια άλλη λύση. Και τελικά φαίνεται να περνάει το χρόνο του ο καθένα στο να βρει τη χρηματοδότηση και όχι στο να κάνει τη δουλειά του σωστά και με αποτελέσματα. Νομίζω ότι με το να μιλάμε μόνο έχουμε χάσει το έργο. Δεν ξέρω πού βρίσκεται το ουσιαστικό εμπόδιο. Και κάτι άλλο σχετικό με, την, ε, με το τοπικό εντοπισμό οι μη κυβερνητικέ οργανώσει δηλαδή θα μπορούσαν απευθεία να έχουν ε, ε, την επαφή και την ε, συνδιαλλαγή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν, δεν το επιτρέπουν όμω οι κανόνες. Ωραία, θα απαντήσω λοιπόν. Αν είναι έτσι, γιατί να μην αλλάξουμε κανόνε. Αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε τα χρήματα σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί. Μόνο, μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με την Ελλάδα, μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί και τα καταφέραμε πολύ καλά και γρήγορα. Χρειάζεται λοιπόν το μέσο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όλα τα άλλα έχουν ε, αναθεωρηθεί. Πρέπει και αυτό να αναθεωρηθεί. Το 96 δεν είναι. Κοιτάω και προς, τους, ε, προς τα μέλη των υπηρεσιών μας να μου το επιβεβαιώσουν. Είναι πολύ παλιό. Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, παραδείγματι. Είδαμε μια γυναίκα η οποία είχε ξεκινήσει ένα εξαιρετικό έργο. Ακριβώς αυτό που χρειαζόταν και την υποστήριξη. Πολύ δύσκολες συνθήκες αλλά είχε χρειαστεί να περάσει μέσα από μια δυτική με κυβερνητική οργάνωση. Και άρα είδαμε κάποιους νεαρούς εκεί, από μια δυτική με κυβερνητική οργάνωση και με τα μπλουζάκια τους κτλ. Δεν είναι λίγο πατερναλιστικό όλο αυτό. Να λέμε μετά, α, η τάδε μη κυβερνητική οργάνωση δαπάνησε τα χρήματα για να κάνουν αυτή τη δουλειά οι ντόπιοι. Δεν πρέπει να αλλάξει. Είχα μια συζήτηση με την Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού και εκεί ακριβώς εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι όταν είναι τόσο δύσκολες συνθήκες και πάμε να δαπανίσουμε χρήματα για να κάνουμε κάτι καλό μπορεί κάποτε να μην πάνε όλα άψογα. Συνήθως καλά πάνε, αλλά δεν δέχονται να υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή μια πρόθεση ε, να αποκλείσουμε κάθε πιθανότητα κινδύνου, να μιλούμε με μηδενικό κίνδυνο. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να εξυπηρετεί βέβαια και το κοινοβούλιο, γιατί είναι ωραίο, κάνει και μεγάλου πηχαίου κύκλου όταν μπορεί να ανακοινώσει τα μεγάλα ποσά που θα αναπάνει. αλλά μετά όταν μπει στην ουσία και στη λεπτομέρεια του τι και πώ, ίσω είναι λιγότερο εμφανέ το αποτέλεσμα. Ξέρουμε βέβαια ότι πάντα υπάρχει και η διαφθορά και τα προβλήματα στη διαχείριση. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε του ανθρώπου αυτού που δουλεύουν σε τόσο δύσκολε συνθήκε. Και σε, σε τέτοιο περιβάλλον ή κλίμα στο οποίο αναφερόμαστε, πρέπει να δεχθούμε ότι πάντα θα υπάρχει κίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, το μέσον δεν έχει αναθεωρηθεί, όπω. είπαμε, έχει σχεδιαστεί για άλλε εποχέ ίσω. Έστω μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι κάτι γίνεται, φτάνουν κάποια χρήματα στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί άλλο είναι να δαπανώνται τα χρήματα και άλλο είναι να φτάνουν τελικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να μην έχουμε τους ενδιάμεσους που τελικά εμποδίζουν τη ροή του χρήματο ε, χάνεται ένα ποσοστό. Υπάρχουν βέβαια μεγάλε μη κυβερνητικέ οργανώσει που κάνουν τη σχετική έρευνα και δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με το πόσο από το κάθε ευρώ που έχει δαπανηθεί σε επίπεδο Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνει ε, στου ανθρώπου που το έχουν ανάγκη στι ε, χώρε αποδέκτε. Αυτό όμω πρέπει να το συστήσουμε, πρέπει να φέρουμε κάποια αλλαγή. Αν δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο, δίνω το λόγο στου ομιλητέ μα. Ρίκ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα μπορούσαμε να περάσουμε ώρες εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη φυσικά. Ας ξεκινήσω αντίστροφα από τις ερωτήσεις της Λίντα. Το μέσο λειτουργεί αρκετά καλά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξουμε το μέσο αλλά λίγη καινοτομία όσον αφορά την τοπική προσαρμογή, τη χρήση τοπικών φορέων και το πρόβλημα, όπως είπατε, έχουμε τις ελεγκτικές αρχές ε, και την όλη τάση ελαχιστοποίησης ή μεταβίβασης των κινδύνων, γιατί αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Οι δωρητές ε, ουσιαστικά ε, μεταβιβάζουν τον κίνδυνο στους μεγάλους φορείς και αυτοί μεταβάζουν τον κίνδυνο στις μικρές, μικαιό, στις τοπικές ΜΚΟ, στην πρώτη γραμμή και αυτό μεταβάζει όλα τα προβλήματα της ε, ε, αβεβαιότητας. Ε, πρέπει να βρούμε τρόπους να κινούμαστε πιο άμεσα. Να χρηματοδοτούμε τις πολύ μικρές ΜΚΟ φυσικά που εργάζονται σε συγκεκριμένες συνθήκες και δεν έχουν της, ε, την όλη δομή παροχής ε, ε, χρηματοδότησης ώστε να λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση που θα μπορούσε να τους δώσει η Κομισιόν οι μεγάλοι δωρητές. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες χρεοκοπίας. Αν κάτι δεν λειτουργήσει, κάποια τραπεζική ασφάλεια για παράδειγμα, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Ψάχνουμε να δούμε δηλαδή οργανισμούς που καλύπτουν γενικά πολλούς τομείς, πολλές ε, έχουμε δει λοιπόν ε, τι έχει γίνει με μικρές ΜΚΟ, με διάφορους φορείς, οπότε θα μπορούσαμε να ε, καταργήσουμε κάποια επίπεδα και αντί να έχουμε 500 μικρούς εταίρους, να έχουμε κάτι πιο ευρύ. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον, για την εταιρική σχέση στο μέλλον αλλά λαμβάνω υπόψη και αυτά που λέτε και για την ε, πολιτική εφαρμογή όσον αφορά τις συμπληρώσεις ε, συμβάσεων, το πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά. Το είπε το υπόθηκε καθαρά. Ποτέ δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, παρότι είχε αυξηθεί το επίπεδο χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, απορροφήθηκαν όλα από τις επιπλέον κρίσεις αμέσως. Διαρκώ λοιπόν κοιτάμε να δούμε πόσα μπορούμε να δώσουμε εδώ ε, προκαταβολή τι θα πάει στο απόθεμα για περίπτωση έκτακτη ανάγκη, τι θα γίνει με τι πολιετής ε, ε, Όλα αυτά κατακαιρματίζονται τρομακτικά. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τα απλουστεύσουμε και να κόψουμε σίγουρα και μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας ε, που αγγίζει και τους εταίρους μας. Αυτά θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στι επόμενε συμφωνίες. Για τα όσα ρώτησε ο κύριος Γκερέρο Σαλώμα για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι σίγουρα η πρόταση είναι να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για το ανθρωπιστικό μέσο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ανάπτυξη. Δεν είναι καλό να έχουμε περισσότερα χρήματα για ανθρωπιστικούς σκοπούς και λιγότερα για αναπτυξιακούς. Ε, η μετάβαση μεταξύ των δύο θα πρέπει να γίνει ομαλά κομμάτι της προτάσης της Κομισιόν είναι να υπάρξει ειδική χρηματοδότηση για ε, βελτίωση της αντοχής, για τιμότητα, για διάφορες παρόμοιες πτυχές. Θα δούμε πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, αλλά προφανώ καλό θα ήταν ε, το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει κάποιε από αυτέ τι ιδέε και να χρηματοδοτήσει επαρκώ κάποιε από αυτέ τι ιδέε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά επί τόπου στους τοπικούς παράγοντες, στους τοπικούς φορείς. Ναι, Πράγματι, όσον αφορά την αντίδραση αντί για την πρόληψη, αυτό ισχύει για τις φυσικές καταστροφές. Νομίζω ότι έχουμε φέρει λίγο καλύτερα αποτελέσματα στα θέματα ε, πρόβλεψης. Κάτι άλλο που λαμβάνουμε όλο και περισσότερο υπόψη μας στον ανθρωπιστικό κλάδο είναι το πώς οι σειράξεις ε, και οι σχετικές δυναμικές ε, επηρεάζουν την ανθρωπιστική απόκριση. Δεν λέμε ότι πάντα πρέπει να έχουμε ειρηνευτική διαδικασία ως στόχο, αλλά αν μπορούμε να συμβάλλουμε μέσω μιας ανθρωπιστικής απόκρισης σε ε, θετική έκβαση και κάποια σύραξη ε, ή σε νωρίτερη ε, λήξη μια σύραξη είναι καλύτερο, είναι πιο αποτελεσματική και να μην συνεχίζουμε να πέφτουμε σε σειράξεις που είναι προβλέψιμες εντελώς όπως έγινε με το Μιανμάρ και το Μπαγκλαντές ε, υπήρχε προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρόνια και παρόλα αυτά συνέβη. Οπότε όταν βλέπουμε κάτι, ε, προβλέπουμε κάτι, να αντιδράμε αρκετά νωρί. Κάτι τελευταίο. Η κυρία Χόιμπουχ ε, και θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ισχύει πράγματι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει ό,τι μπορεί. Γι' αυτό το λόγο, αυτός είναι ένας από τους λόγους, ε, ε, έχουμε κάτι τόσο κατακαιρματισμένο ε, και μετά προσθέτουμε πράγματα, συμπληρώνουμε πράγματα ή χρειάζεται να ξεκινάμε από την αρχή. Θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα πράγματι, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πολλοί από τους νέους δωρητές ε, έχουν μεγάλα μέσα και τελικά δεν καταφέρνουν ή καταφέρνουν πολύ αργά ή χρειάζεται πολύ ε, μεγάλος ε, πρόορος προγραμματισμός για κομμάτια μόνο μιας κρίσης ή για συγκεκριμένους εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει ουσιαστικά να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και μετά αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και από την αναπτυξιακή πτυχή φυσικά ε, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά ώστε κάποια χρήματα να δοθούν εκεί, πώς μπορούν να δαπανηθούν εκεί σε σχέση με την ανθρωπιστική πλευρά. Ε, να δείξουμε δηλαδή λίγο μεγαλύτερη ευελιξία. Ευχαριστώ, θα σταματήσω εδώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουγλό. Thank you and thank you very much for the different uh, Σας ευχαριστώ ε, και για τα σχόλιά σας. Δεν έχω ε, ερώτηση εγώ να απαντήσω που να μου έχει γίνει άμεσα σε μένα. Ε, για την επιτόπου διαχείριση και την αξιολόγηση και την αναθεώρηση ε, της πολιτικής. Υπάρχουν τα σωστά εργαλεία, θα πρέπει να βρεθεί ένας καινοτόμος τρόπος να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της μεγάλης συμφωνίας αυτής, Grand Bargain. Αλλά αυτό εμείς ε, που θέλουμε είναι απλούστευση, χωρίς απλοποίηση των διαδικασιών. Ε, δεν υπάρχει ε, τρόπος και λόγος να γίνεται επιτόπου η διαχείριση αυτών των διαδικασιών από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν έχουν ούτε τους πόρους, ούτε τα μέσα, ούτε τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Grand Bargain δεν είναι απλώς ε, η μετατόπιση και η νέα φιλοσοφία ότι δίνουμε χρήματα επιτόπου στις οργανώσεις, αλλά αλλάζουμε τελείως και νοοτροπία και διαχείριση. Και ε, τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει ε, να ενστερνιστούν αυτή την προσπάθεια και να την εντάξουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και η φωνή των οργανώσεων αυτών θα πρέπει να ε, ακούγεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, άλλοι αρμόδιοι φορείς για την ανθρωπιστική βοήθεια πιστεύουν και πιέζουν προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, η ε, αναπτυξιακή κοινότητα θα πρέπει όλα αυτά να τα υιοθετήσει Δεν πρόκειται για άμεση έκτακτη βοήθεια. Και στον υπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό κονδύλι για τη βοήθεια στη δημιουργία ανάπτυξης ε, ικανοτήτων επιτόπου ακριβώς για τις οργανώσεις για να μπορούν να εφαρμόζουν όλα αυτά τα κριτήρια που καλούμαστε να θα υλοποιήσουμε. Υπάρχουν διάφορα στρώματα τώρα στην αρχιτεκτονική λήψη απόφαση και χρηματοδότηση. Συμφωνώ, αλλά πρώτα να κοιτάξουμε γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα στρώματα. in, ε, Ορισμένοι από τους εταίρους αυτούς σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι πραγματικά πολύτιμοι και προσθέτουν αξία στην όλη διαδικασία. Ορισμένα από τα μέλη του δικτύου Voice ε, έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν σε μια εταιρική σχέση, έχουν στείλει ένα χάρτη για την αλλαγή ε, και είναι πάρα πολύ ε, σοβαρή η συμμετοχή και η δέσμευση. Υπάρχουν και άλλες οργανώσεις ανθρωπιστικές όπως είναι η Κάριτας που βοηθούν πάρα πολύ στη δημιουργία ικανοτήτων των τόπιων εταίρων των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας επιτόπου. δεν είναι ένα το στρώμα, ας πούμε, ε, μπορεί σε μία σύμβαση να φαίνεται ότι είναι ένα ο εταίρος, αλλά είναι πολύ πιο περίπλοκη η εικόνα. Αυτά. Προσβλέπουμε στο επόμενο διάστημα να δούμε τι θα προκύψει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Στη νέα διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο FBI. Ένα ζήτημα που γενικά αντιμετωπίζουμε σε διάφορους τομείς πολιτικής Πώς θα δώσουμε φωνή δηλαδή στον πολίτη. Πώς θα μπορέσει αυτό που θα προσφέρουμε να αλλάξει πραγματικά τη, ζωή του. Γιατί μπορεί να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις και να νομίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο. Αλλά στην πραγματικότητα πώς βοηθούμε. Και σε άλλους τομείς δημόσιας ε, πολιτικής και παρέμβασης υπάρχουν μοντέλα που μάλιστα και εγώ στην προηγούμενη μου σταδιοδρομία είχα ε, αναπτύξει. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που μπορεί να έχει ας πούμε, η κάρτα ως οργάνωση, να παίρνει το μεγάλο ποσό και μετά να το κόβει σε πιο μικρά και να το χορηγεί στον, ε, σε μικρότερες ομάδες ή σε μεμονωμένους πολίτες. Αλλά όπως και να έχει και με όλη την καλή δουλειά που μπορεί να γίνεται εκεί, τέσσερα χρόνια είμαι πρόεδρος εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης και διαρκώς το ίδιο πρόβλημα ακούμε και έχουμε την εντύπωση ότι οι χορηγοί πολλές φορές δεν ακούν, δεν αφουγκράζονται αυτό που χρειάζεται. Πολλές φορές με ένα πολύ πολύ μικρό ποσό μπορεί να εξασφαλίσουμε τεράστιες αλλαγές. Μέσα περιπτώσει δεν ξέρω πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Το FPR θέλετε λίγο να μας ενημερώσετε έστω για το Χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ευχαριστώ. Πρόκειται για συζητήσει κανονικά μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των διαφορών εταίρων. Φυσικά, όπω είπατε και εσεί, έχει να κάνει με τη βελτίωση τη ε, βοήθεια πιο, με πιο αποτελεσματική βοήθεια, με πιο μεγάλο αντίκτυπο είναι κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε έτοιμο για το τέλος του 2019 και νομίζω ότι οπωσδήποτε και ε, είναι σύμφωνο με τα όσα έχει στήσει μάλιστα το, το συντρέχουσα στην τρέχουσα θητεία του και σύνθεσή του που ακόμα θα είναι ε, αλλά και με το πολιτισμικό πλαίσιο. Καλώς ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τις ομιλήτριες για την ενημέρωση. Okay, we have votes coming up, so we're going to move swiftly. Έπονται ψηφοφορίες. Ας επιταχύνουμε λοιπόν λίγο. Η Σύμβολη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνιστικό Χαρακτήρα μα του ΙΕ σχετικά με τι διεθνικέ εταιρείε και άλλε επιχειρήσει με διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχω αναλάβει εγώ ω πρόεδρο τη Επιτροπή και εδώ έχουμε να κάνουμε με δεσμευτικό μέσον για τις διεθνικές ε, συνεργασίες, ε, συνεργασίες του 2014 αποφάσισαν ο Βουλίο Ασφαλείας των ΗΠΑ να θεσπίσει την ε, διακρατική ομάδα εργασίας IGAG για την θέσπιση ενός μέσου που θα παρακολουθούσε με βάση το Διεθνές Δίκαιο τις εργασίες των διεθνικών οργανώσεων. Έχει συνέλθει τρεις φορές. Η τέταρτη σύνοδος προβλέπεται για τον Οκτώβριο της, Επιτροπής, ε, της ομάδας αυτής εργασία, εργασίας, την οποία εμείς παρακολουθούμε εξ αρχής στις δραστηριότητές της και θέλαμε αυτή η συζήτηση να συνοδευτεί από προφορική ερώτηση και ψήφισμα πριν από την προσεχή σύνοδο του Οκτωβρίου. Ε, μάλλον η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει ε, στις θέσεις, σε θέσεις δικές της, επομένως έχει ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα το τι κάνουμε εμείς. Ε, τώρα θα πρέπει να ε, δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε αυτό το ψήφισμα για να είναι έτοιμο για ψηφοφορία των, ε, για συζήτηση μάλλον τον Ιούλιο. Δίνουμε ήδη την ευκαιρία για τις τροπολογίες 186 είναι οι τροπολογίες που έχουν μέχρι τώρα κατατεθεί. Και η, Επιτροπή, η Υποεπιτροπή των ανθρωπινών Δικαιωμάτων έχει κάνει προτάσεις. Θα καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές γενικά. Συζητούμε τα θέματα αυτά. Ο Μπόγκταν Βέντα έχει το λόγο όμως πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, έχουμε το προφορική ερώτηση για το δεσμευτικό μέσο των εθνών και τη διακρατική συνεργασία. Εγώ ως και όδης της ομάδας μου υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να απευθύνουμε ερώτημα προς την Επιτροπή και να λάβουμε και καμιά απάντηση. Ωστόσο, εμείς πρέπει, έχουμε ξεκινήσει το ψήφισμα χωρίς να περιμένουμε την απάντηση της Κομισιόν. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες και ελπίζουμε ότι στη διαπραγμάτευση με τι άλλες ομάδες θα καταφέρουμε να βρούμε κοινό τόπο παρότι κάποια από τα θέματα του ψηφίσματος είναι σημαντικά κατά την άποψή μου το θέμα αυτό είναι περισσότερο αρμοδιότητα τη ΣΥΝΤΑ και όχι δικό μας. Όσον αφορά το μέσο, ε, το μέσο. Αρκετά κράτη ναι, έχουν δεχθεί το δικό τους μερίδιο για την προσβάση στην αγορά. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Πολλές χώρες δεν συμμετέχουν στην επόμενη ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, όταν θα κάνουμε έκκληση για ε, υποχρεωτικές απαιτήσει για τις ευρωπαϊκές εταιρείε ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δημιουργεί ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές χώρες Οπότε είναι σημαντικό να εγγυηθούμε ότι όλες οι μορφές ε, επιχειρηματικότητας παγκοσμίω θα συμπεριληφθούν επαρκώς ε, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τζούτιθ, θέλατε το λόγο, Τζούτιθ. Ναι, πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα στείλουμε αυτή την προφορική ερώτηση και ελπίζω να ψηφίσουμε και κάποιο ψήφισμα με σαφή στάση να προκύψει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οποία θα παροτρύνουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν να δείξουν θετική στάση προς ένα παγκόσμιο δεσμευτικό μέσο. Διότι μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ανέλαβαν οι χώρες στη Γενέβη στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτό το θέμα ε, και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αρχικά δεν ε, είχαν καθόλου θετική στάση. Αντιθέτω, προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν ουσιαστικά την ε, διαδικασία, να την κάνουν να και πιστεύω κάποια κράτη-μέλη έχουν πει ότι είναι το υποστηρίζουν και πιστεύω ότι θα μας βοηθούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δουν το πράγμα λίγο πιο θετικά. Στο μεταξύ, διαπραγματευόμαστε εμπορικές συμφωνίες με συστήματα επίλυσης διαφορών για μεγάλες επιχείρησεις αλλά δυσκολευόμαστε να δώσουμε σε πολίτες ε, το δικαίωμα σε τρίτες χώρες ε, να έχουν κάποια πρόσβαση ένδικα μέσα σε περίπτωση που κάτι διακυβεύεται για αυτούς. Ε, χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Κρίμα που διστάζουν οι φίλοι μας από την ίντα. Αλλά το προωθήσουμε ας και έχουμε μια καλή ψηφοφορία ε, στην ε, Ολομέλεια πριν από τη Σύνοδο του Οκτωβρίου. Ευχαριστώ η κυρία Χάουτελα. Αλλά προηγουμένως η Λόλα Σάντσετ. Ευχαριστώ πολύ Λίντα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σου εργασία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή βάση η συμβιβασμοί που προτείνεις για να προχωρήσουμε και πραγματικά μπορούμε να ανταποκριθούμε στο βασικό μας στόχο που είναι να ε, διαβιβάσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την τεχνογνωσία μας, αλλά και την υποχρέωσή μας να εκπροσωπούμε τη φωνή των πολιτών και να φτάσει αυτό μέχρι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ε, για να σχολιάσω κάτι πάρα πολύ σύντομα, μερικά πράγματα που είδα σε σχέση με τις τροπολογίες του κειμένου, εγώ δεν κουράζομαι να λέω ότι αυτό το μέσο είναι απολύτως συμβατό με πάρα πολλά άλλα που έχουμε. Ας πούμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τις εθνικές νομοθεσίες που έχουν ε, εγκρίνει κάποια θαραλέα κράτη προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα Με εκπλήσουν οι τροπολογίες κάποιων συναδέλφων που λες και ντρέπονται ε, να ε, μιλήσουν για κάποια πράγματα που είναι προφανή και αυτονόητα. Ότι θα πρέπει να κυριαρχούν τα ανθρώπινα δικαιώματα επί διαφόρων ε, συμφερόντων. Και κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να απορριφθούν τέτοιε τροπολογίε που ακριβώ αυτό δηλώνουν, ότι είναι απόλυτη κυριαρχία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οχτώ φορέ έχουμε πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα οι εκθέσεις ότι υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης να είναι επικοδομητική στη τους και όχι καταστροφική όπως μέχρι τώρα. Είναι επίδειξη και ένδειξη οριμότητας ε, αυτό και πολιτική σύνεση. Υπάρχουν πολλά κενά για τη δικαιοσύνη και την επανόρθωση και την αποζημίωση στην οποία έχει δικαίωμα το κάθε ε, άνθρωπος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε ακόμα ένας φορέας, ε, ο πρωταγωνιστής ε, για να κάνουμε προτάσεις αυτό το δεσμευτικό σχέδιο κειμένου. Και όχι απλώς επειδή συμπίπτει με τις δικές μας αρχές και αξίες, αλλά γιατί είναι και ο ίδιο ο λόγος ύπαρξης ε, του θεσμικού μας οργάνου και γιατί χρειαζόμαστε ένα σαφέ, ενιαίο και χρήσιμο ε, νομικό πλαίσιο ε, που να καλύπτει τα κενά. Μπορούμε λοιπόν να εργαστούμε με βάση αυτό το κείμενο και ελπίζω να έχουμε μια ευρεία συνένεση όπου θα προέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα πέραν οποιοδήποτε άλλον. Κυρία Χάουταλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τη σημασία αυτής της διαδικασίας που έχουμε στο Κοινοβουλίο με τις τρεις επιτροπές με την, εξωτερική υπηρεσία, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή, όλη αυτή η δουλειά που έγινε. Ήταν πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή διστάζουν είναι ότι αυτή η, διαδικασία, αυτή η πρωτοβουλία αρχικά αφορούσε διεθνείς εταιρείε ενώ αν κοιτάξουμε την παγκόσμια λυσίδα αξίας δεν πρέπει να αποκλείονται οι εγχώριες εταιρείε. γιατί τότε ε, χάνεται η διαφάνεια στην αλυσίδα της προμήθειας και ταυτόχρονα όλη αυτή η ιδέα δεν έρχεται σε αντίθεση με τη λεγόμενη δεσμευτική συνθήκη, γιατί μπορούν να υπάρχουν ε, άλλοι όροι, όπως η ιδέους επιμέλεια, όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, και προϋποθέσεις που οδηγούν σε παρέκκληση από τα όσα έχει συμφωνήσει ο Ρωσμός των Μοναδινών. Πάντως τώρα έχει λάβει εντολή για την πραγμάτευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοδομητικός ή μη είναι κάποιο μόνο όταν έχει μια εντολή διαπραγματεύση. Μόνο από εδώ και μπρος λοιπόν μπορεί να γίνει. Και επίση για του συναδέλφου και σε σχέση με την ίντα στην οποία επίση είμαι μέλο. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουν τη σημασία αυτή τη πρωτοβουλία. Και ελπίζω ότι θα μπουν και αυτοί στο χώρο. Καλώς. Λοιπόν, έχουμε εδώ την Επιτροπή την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που είναι αρμόδια κατ' ουσίαν θα έλεγα καθήλεν. Ο Μάρκ Τζακομίνη είναι εδώ για να μας πει ποιο είναι αυτό το ιστορικό της εντολή τι έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και επιτρέψτε μου καταρχάς να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με εταίρου από διάφορες περιφέρειες για την υλοποίηση της πρότασης του πλαισίου που υπενθυμίζει βεβαίως διαρκώς την υποχρέωση για τήρηση των νομικά όρων. Η υποχρέωση για κάλυψη των κενών. Χαίρομαι διτέρως που η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες για ανταλλαγή, για πρόοδο. 17 Μαΐου, παραδείγματι, είχαμε τις διαβουλεύσεις της ομάδας, στην οποία λάβαμε μέρος ιδέους επιμέλεια αλλά και άλλες πρακτικές έχουν σημασία ως προς αυτό και έχουμε προτάσεις προς, τις, ε, προς τα προξενία με τα ένδικα βοήθηματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε επίσης ε, πρόσβαση στα ένδικα βοηθήματα που προτείνουμε σε ένα έγγραφο του Συμβούλου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα δει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκ τούτου υποστηρίζει πλήρως το ψήφισμα με τις προτάσεις της ε, Αργεντινής, της Γκάνας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πρόσβαση στα ένδικα βοηθήματα. Είναι πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το στηρίξει για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των στόχων των ΗΠΑ για το νομοθέτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διστάζει ως προς... Η Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει και σκέφτεται λίγο εάν χρειάζεται ένα νέο νομοθέτημα, χωρίς να αντιτίθεται σε αυτό και έχουμε άλλωστε επικοδομητικά συζητήσεις. τις τελευταία συνόδο της διακυβερνητικής ομάδας ήμασταν μάλιστα και πιο δραστήρια αντιπροσωπεία ζητώντα διευκρινήσεις και δεν δεχόμαστε είπε ότι δεν είχε συμμετοχή στη διαδικασία η πλευρά μας, ούτε ότι ήταν καταστροφική αντί για επικοδομητική συμμετοχή αυτή. 14 Ιουνίου του 2018 είχα μια τελευταία σύνοδο, στην οποία μόνο τε, ο λίγα κράτη ε, μίλησαν για την ουσία και πιστεύουμε ότι πρέπει η διαδικασία να προχωρήσει, να λυθούν τα διαδικαστικά ζητήματα. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα στα δικονομικά ζητήματα κατά τρόπο αντικειμενικό. Ενδεχομένως και με ψήφισμα από το Συμβούλιο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και ενδεχομένως και με μια παραπομπή στη συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Με αυτή τη μορφή ή με κάποια άλλη. Οπωσδήποτε χρειάζεται σαφές χρονοδιάγραμμα και ορόσημα με βάση και τις παγιωμένες τακτικές. Ο πρώην πρέσβης Λόγκ έχει ζητήσει να γίνει η αναφορά στην Τετάρτη Σύνοδο 14, 15 Οκτωβρίου με το Εκουαδόρ στην σύνταξη, αλλά δεν το έχουμε δει το κείμενο ακόμα. Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε για τις καθυστερήσεις, για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες, οι κυβερνητικές οργανώσεις, και διάφοροι άλλοι φορείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την απουσία δεσμευτικών κανόνων. Είναι σαφές πως είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι χρειάζεται να ξέρουμε τι είδους πολιτική δέσμευση χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα και, την, ε, και να δώσουμε προστασία στα θύματα των καταχρήσεων. Έχουμε συζητήσει με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ενημερώνουμε τους συντονιστές στην ομάδα. Πρόκειται για διάλογο που κρατάει αρκετά χρόνια και βέβαια εμπλέκει σε συνομιλίες στην Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία και τα κράτη-μέλη, ορισμένα από τα οποία έχουν αναλάβει και την πρωτοβουλία για επαφές σε διεθνέ επίπεδο. Πρωτοβουλία, πρωτοβουλίες που ξεπερνούν οτιδήποτε άλλο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο Μιλούμε και για νομοθεσία και σε ευρωπαϊκό και σε κρατικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των στόχων. Έχουμε επαφές και προγραμματίσει σύνοδο με εκπροσώπους διαφόρων φορέων όπως συνδικαλιστικά σωματεία, με κυβερνητικέ οργανώσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις για να δούμε στοιχεία της πρακτικής υλοποίησης. θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προσπάθειες για εφικτές και βιώσιμες λύσεις. Σε σχέση με την εντολή, πρώτα χρειάζεται σχέδιο συνθήκης, σύμβασης και μετά θα καταθέσουμε τις προτάσεις και τις θέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δουλειά ακόμα για να έχουμε τη συμμετοχή και των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, χρειάζεται τη συμμετοχή των κρατών μελών. Λοιπόν, συνάδελφοι, προτείνω να τα μείνουμε εδώ, να υιοθετήσουμε το, την προφορική ερώτηση και να ξαναδούμε το ζήτημα τον Ιούλιο όταν θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Πάμε στο σημείο 9 και θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία είναι εύκολη. Ψηφίζουμε για την προφορική ερώτηση με ονομαστική ψηφοφορία για τη δεσμευτικού χαρακτήρα μέσου που μόλις συζητήσαμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Where's the screen? Uh, I yeah. Has everyone voted? Ψήφισαν όλοι. Ναι. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Υιοθετήθηκε η προφορική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Πάμε τώρα στο σημείο 10. Εκτός μικροφώνου η πρόεδρος. Δυστυχώς δεν ακούμε. Η πρόεδρος είναι εκτός μικροφώνου, δεν ακούμε. 10. Σημείο 10. Διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στι αναπτυσσόμενε χώρε, η περίπτωση των δασών. Είναι μεγάλη η ψηφοφορία αυτή. Πρέπει να ψηφίσουμε τι δικέ μα τροπολογίε και τι τροπολογίε μελών άλλων επιτροπών. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ, Λίντα. Ήταν αρκετά επικοδομητική και συνενετική η διαδικασία. Πιστεύω ότι όλες οι τροπολογίες αφορούσαν διευκρίνηση λεπτομεριών, προσθήκη κάποιων πτυχών που έλειπαν. Δεν υπήρξε πραγματική διαφωνία. ή ελάχιστες σε όλες αυτές τις τροπολογίες. Ε, ήταν εύκολο να βγάλουμε και τις ε, συμβαστικές. Ε, ήταν μεγάλη έκθεση. Πιστεύω οι συνάδελφοι θα παραμείνουν ικανοποιημένοι. Τώρα αναμένουμε η Επιτροπή να προχωρήσει σε, σε κανονική διαβούλευση ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική για την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συντάκτες της Επιτροπής ΕΜΒΗ, την κυρία Καμιάνσκα και την κυρία Αρένα από την Ίντα, διότι πραγματικά συμπλήρωσε η δουλειά της μίας τη δουλειά της άλλης. Ε, ελπίζω λοιπόν έτσι να επιτύχουμε ένα ε, έγγραφο αποτελεσματικό, δυνατό και πρόεδρος και φυσικά και σχετίζεται με το προηγούμενο σημείο κατά πολλούς τρόπους η, η δασοκομεία. Οπότε, Πάμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με τη συμβαστική 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 169 υπέρ κατά εποχές Να ελέγξουμε την 169. Νομίζω εγκρίνεται. Να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV32 υπέρ κα... καταπίπτει, συγγνώμη. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 86 ξεκινάει η ψηφοφορία νομίζω θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται αλλά όχι όσο μεγάλη πλειοψηφία θέλαμε ε, αρκετή συμβεστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV21 υπέρ να ψηφίσουμε unblock είναι δύο μόνο μέχρι να βρούμε άκρη να τις κάνουμε από για τις MV και ίντα μέχρι την MV23 να τις δούμε αν μπλοκ όλες ωραία. ωραία όλο αυτό το μπλοκ λοιπόν κατά αποχές εγκρίνονται όλες ευχαριστώ πολύ 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, συγγνώμη, απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα απορρίπτεται καταπίπτει διότι απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 112, άρχεται ε, η ψηφοφορία, νομίζω απορρίπτεται. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. MV25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είτε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα της 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ίδιο για την 137 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 έχει αποσυρθεί 140 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Λοιπόν, 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 151 έρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται νομίζω ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται οι ίδιες ε, πλειοψηφίες είναι τα 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV28 υπέρ κατά είναι σε δύο τμήματα Πρώτο τμήμα της ΕΜΒΙ 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την συμβιβαστική 26 άρχιτη ψηφοφορία. Η συμβαστική 26 ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Ναι, ίδια πλειοψηφία. 13-8. MV 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει unblock η 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 Α, συγγνώμη, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Είναι 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, πάμε σε τηλεολογικές σκέψεις. Ε, πήγαμε γρήγορα. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να δούμε Έχουμε μόνο λίγε. 70 ε. υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 71 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 19 καταπίπτει, 63 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Πάμε μετά block για τι επόμενε 72 μέχρι 30 υπέρ. Α, δεν θέλετε, 72 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές να την ξανακάνουμε λοιπόν 35 ξανά 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται να ελέγξουμε τη 36 άρχεται η ψηφοφορία Is everybody, ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ελέγξουμε τη 43, ναι, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 43. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 45 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα καταπίπτει λοιπόν 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβεστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 καλύπτεται από τη συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 και 59 η 58 απορριφθήκε την 60 δεν την ψηφίζουμε, η 59 εγκρίθηκε. Η 60 καλύπτει από την άλλη τροπολογία. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε αιτιολογικές αναφορές, να τις δούμε αυτές σαν μπλοκ όχι. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε είπατε.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 11. Να ξαναδούμε την 11. Συγγνώμη, δικό μου λάθο λέει η πρόεδρος. Είμαι πολύ γρήγορα. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται νομίζω να ελέγξουμε την 11. Άρχεται ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε επί του συνόλου της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Χάτελα. Ομόφωνη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Πάμε στο 11. Φεύγει ο κόσμος. Αυτή που φεύγεται παρακαλώ αποχωρείτε ησύχω. Λοιπόν, πάμε στην ώρα των ερωτήσεων. Έχουμε την ερώτηση του Ερίκε Κεραίρο προ την Κομισιόν. Δεν θα διαβάσω. Ουσιαστικά αφορά το πώ η ΕΚΟ... Συγγνώμη, ησυχία. Όσοι φεύγετε στην ώρα των ερωτήσεων, επειδή θέλουμε να μιλήσουμε. Αν θέλετε εσεί να μιλήσετε, μιλήστε εκτό τη αίθουσα, γιατί πάμε στο σημείο 11, ώρα των ερωτήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αφορά τη χρηματοδότηση των προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας. Και ζητάμε από την ΕΚΟ να μας πει τι κάνουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά από τις περικοπές στη ροή χρηματοδότησης τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ από την ΕΚΟ για να απαντήσει. Παρακαλώ, οπότε έχω το όνομά σας, συστηθείτε παρακαλώ. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τη Λόριδα της Γάζας και την ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΕΚΟ. Αν δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση, παρακαλώ βγείτε από την αίθουσα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Βελενσιάνα Περνάρτη από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Ε, είμαι επικεφαλής της ομάδας για το ε, Ιράκ και την Παλαιστίνη. Γενικά σχόλια για να θέσουμε το πλαίσιο και μετά θα περάσω μέσω στην απάντηση. Ανησυχούμε βαθύτατα για τις επανελεινόμενες ε, συγκρούσεις που ξεκίνησαν από τις 30 Μαρτίου και συνεχίζονται μέχρι τον Ιούνιο στα σύνορα με τη Γάζα. Όπως γνωρίζετε αυξάνεται ο ρυθμός των θυμάτων. Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για 135 νεκρούς και πάνω από 14.600 τραυματίες. Και δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία της περασμένης Παρασκευής, αλλά με βάση ανεπίσημα στοιχεία φέρουν 200 ε, επιπλέον ε, τραυματίες. Υπάρχουν επίγουσες ανάγκες ε, και αν δεν αντιμετωπιστούν θα έχουν επιπτώσεις μέσω μακροπρόθεσμα για το σύστημα υγείας στη Γάζα και όλο τον άμαχο πληθυσμό. Η κατάσταση ήταν έτσι κι αλλιώς ε, δεινή με μια οικονομία μετά από 11 χρόνια ε, αποκλεισμού. Ε, το νερό, η αποχέτευση και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι περιορισμένα. Ο κόσμος ζει στη φτώχεια, στην ανεργία και χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή λοιπόν η αποανάπτυξη θα πρέπει να αντιστραφεί υπάρχει και κρίση ρευστότητα στη Γάζα λόγω και μείωση της χρηματοδότησης επειδή δεν ε, μπορούν οι αρμόδιοι φορείς για την ανθρωπιστική βοήθεια να ανταποκριθούν. Απαντώ στην ερώτησή σας, τι ε, βήματα έχει ε, σχεδιάσει η ΕΚΟ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η αρχική χρηματοδότηση που είχαμε προβλέψει ήταν 21 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 70% περίπου έχουν προσημειωθεί για τη Γάζα και έχουν συναυθεί και αντίστοιχε συμβάσει. Το τελευταίο δίμηνο έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Ε, κάθε εβδομάδα συγκρούσει, Και έχουμε και περιορισμένες ε, δυνατότητες ε, δράσης λόγω του αποκλεισμού της πόλης της Γάζας και της, των διακοπών στο ρεύμα. Έχουν ε, αποφασιστεί 3 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ως ανθρωπιστική βοήθεια ε, σε τομείς όπως είναι υγεία και αποχέτευση. Καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών για την προετοιμασία για έκταξη ανάγκες, τη στέγαση, την υγεία και την αποχέτευση. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και οι εταίροι οργανώσεις επιτόπου παρακολουθούν την κατάσταση. Πάνω από 270 εκατομμύρια ε, ευρώ έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας. Ρωτάτε, ε, ρωτάτε αν θα υπάρχει ειδική χρηματοδότησης. Σας είπα, έχουν κινητοποιηθεί το Μάιο 3 εκατομμύρια ευρώ. Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά για να δούμε πώς θα μπορέσουμε ευέλικτα να απαντήσουμε σε περίπτωση που υπάρξουν επιπλέον ανάγκες. Βεβαίως σκεφτόμαστε ε, να κινητοποιήσουμε και άλλα κονδύλια. Ρωτάτε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τον ιστορικό μηχανισμό πιο ε, ευέλικτο για να συνδεθεί η αναπτυξιακή με την ανθρωπιστική βοήθεια. Επειδή τραβάει σε μάκρο αυτή η κατάσταση και λόγω των ε, πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων θα πρέπει να συνδεθεί η ανθρωπιστική με την αναπτυξιακή βοήθεια ε, στην Παλαιστίνη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να πιάνει τόπο η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα να είναι βιώσιμη η λύση των δύο κρατών. Οι υπηρεσίε μας συνεργάζονται το τελευταίο διάστημα όλο και πιο στενά, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τι πιο ευάλωτες οικογένειε στη Γάζα που εξαρτώνται πάρα πολύ από τη βοήθεια και αυξάνεται η φτώχεια και η ανεργία. προ το σκοπό αυτό σε επίπεδο διευθυντών το Φεβρουάριο διοργανώθηκε αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ, ΝΙΑΡ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την ούνρα που έχει πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αυτό έχει επίπτωση στην καθημερινή ζωή ευάλωτων Παλαιστινίων ε, προσφύγων στη γύρω περιοχή και στην ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ και στο Λίβανο, την Ιορδανία και αλλού αυξάνονται οι εντάσεις και μέσα στην κοινότητα των προσφύγων την ίδια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιταχύνει έτσι ώστε βραχυπρόθεσμα να καταβληθούν τα κονδύλια 82 εκατομμύρια ευρώ από την ε, Γενική Διεύθυνση ε, ΝΙΑΡ. 100% βαρύ σε χρηματοδότηση. Επιπλέον έκτακτο μέτρο. 50 εκατομμύρια πρόγραμμα για τους Παλαιστίνιους ε, πρόσφυγες και τους πρόσφυγες από τη Συρία στο Λίβανο και την Ιορδανία. Και 3 εκατομμύρια για συνεχιζόμενα προγράμματα. Άρα η ευρωπαϊκή γειτονία χρηματοδοτεί με 100 εκατομμύρια. Και η Ούρα υποστηρίζει προγράμματα στη Γάζα με παροχή στέγης. Το 2018 εμείς θα στηρίξουμε τις δράσεις της ώρα για την υγεία με 2 εκατομμύρια ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ε, σταθερός παραστάτης και προβλέψιμος εταίρος για την ώρα. Το ε, Ιούνιο του 2017 υπογράψαμε μια κοινή δήλωση με την ούρα για την στήριξή μας και τη χρηματοδότηση προς την ούρα. Και αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη ότι ε, και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε στο πλευρά τους. Μέχρι τώρα για το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει 106 εκατομμύρια στην ώρα. Ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν μεγαλύτεροι δωρητές και πάροχοι βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αυξήσουμε ε, ιδιαίτερα τις απώλειες που έχουν από τις Ηνωμένε Πολιτείες. αλλά προσπαθούμε να βρούμε και άλλους δωρητές και να τους ενθαρρύνουμε για να συνεχιστεί ή να αυξηθεί η πρικοδότηση προς την ε, ούρα. Ο Ενρίκε Γκερέρο, ο συντάκτης της ερώτησης. Καταρχάς, θα ήθελα όχι απλώς να ευχαριστήσω ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση, αλλά και να τη συγχαρώ, διότι ήταν ευρύτατη, εκτενέστατη, εμπεριστατωμένη, με πολλές πληροφορίες, πάρα πολύ κατανοητή που δεν συμβαίνει πάντα όταν κάνουμε ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση και σας ευχαριστώ πολύ. Η απάντησή σας ήταν ε, εκτενέστατη και πολύ εμπεριστατωμένη. Ε, πώς προέκυψε αυτή η ερώτηση. Είχα μια συνάντηση ως εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια με εκπροσώπους τη ΟΥΡΑ στις Βρυξέλλες που μου είπαν, όπως είπε και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι μετά τις τελευταίες συγκρούσεις είχαμε μέχρι 14.000 τραυματίας ε, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ε, είχαν κατάγματα, και ε, χρειαζόντουσαν χειρουργείο. Άρα κατέρευσε το σύστημα υγείας της Γάζα. Οπότε είπαν ότι ήταν επίγουσα η ανάγκη να βρουν 10 εκατομμύρια ευρώ για το, επόμενο δίμηνο. Η συνεδρία σε αυτή ήταν πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Γάζα, στην οποία δεν θέλω να μπω τώρα, την ξέρετε, ε, τα πολιτικά και τα λοιπά, και εδώ και χρόνο μια κρίση η περιοχή, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και πάρα πολύ από την τιμωρία εντό εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπομορφή μείωσης ή περικοπών της βοήθειας στην ώρα. Λαμβάνουμε υπόψη ότι η Λωρίδα της Γάζας ζει μια κατάσταση ανοιχτής φυλακής. Υπαίθριας δηλαδή, όπου δύο εκατομμύρια ε, άνθρωποι ε, ζουν ε, υπό πάρα πολύ δεινές συνθήκες και χρειάζονται οπωσδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την ευθύνη να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ε, με τη συμπεριφορά αυτή που είχαν και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ανάγκες στο άμεσο μέλλον και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε μια μικρή ενημέρωση για το πώς συνδέεται τώρα η ώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανταποκριθείτε σε αυτές τις άμεσες ανάγκες και τα αιτήματα ε, από την επιδείνωση της κατάστασης. Um, Δεν ζήτησε κανείς άλλος το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Sorry, Annie Leeds asked for Συγγνώμη, Annie Leeds, ε, ε, είδα. E e. Οι διερμηνεί σα ενημερώνουν ότι βρισκόμαστε στην 21η μέρα των κινητοποιήσεων διαμαρτυρία και η διοίκηση παραμένει μετακίνητη. Ύστερα από 8 μήνε διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Προσωπικού, ο Γενικό Γραμματέα αντιθέτω κλείνει τη στάση του και κατά συνέπεια δεν δίνουμε καμία παράταση του ωραρίου και σταματούμε εδώ. in the region, uh, to stress and to get more financial support towards UNRWA. Did that succeed? Did anything happen there as well? Thank you.